Καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλωσορίζω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάριο Ντράγκη. Είναι ο δεύτερος νομισματικός διάλογος που λαμβάνει η χώρα το 2016. Κατά τύχη, η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει η χώρα πολύ σύντομα μετά την απόφαση μες της οποίας το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές κατά του προγράμματος ε, συναλλαγών, νομισματικών συναλλαγών της ΕΚΤ. Χαιρόμαστε που το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφαση του ΔΕΚ του 2015 που λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι εντός της εντολής της ΕΚΤ. Πολύ καλές ειδήσει που ήρθαν πολύ έγκαιρα και επίκαιρε. Στη συνεδρίαση ο πρόεδρος Ντράγκη θα παρουσιάσει τις προοπτικές της ΕΚΤ για οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις, ε, όπως γνωρίζουμε, υπό το φως της αυξήσεως του κινδύνου αντιστροφής ανάπτυξης και της μικρής δυναμικής της πληθωριστικής του ευρώ, στις 10 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε σημαντικές αποφάσεις, ούτως ώστε να χαλαρώσει περισσότερο τη στάση τη νομισματική όσον αφορά τα επιτόκια, την επέκταση της μηνίας αγορά σύμφωνα με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, συμπερίληψη της αγοράς ε, εταιριών του σχετικού προγράμματος και άλλη μια σειρά μέτρων που θα ξεκινήσουν τα μέτρα από αύριο. Η ΕΚΤ συνεχίζει να χαλαρώνει το κόστος των πιστώσεων και συμβάλλει στην ενίσχυση της δημιουργίας πιστώσεων. Θα αναφερθεί στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος της ΕΚΤ, ο κ και πώς ε, αυτό το πρόγραμμα επηρεάζει την ανάπτυξη, πώς επηρεάζει τις επενδύσεις. Πιστεύω θα αναπτυχθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες για τις αρνητικές συνέπειες των παρόντων αρνητικών επιτοκίων που επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία του τραπεζικού τομέα ανάμεσα στις διάφορες μελέτες που παραλάβαμε προετοιμάζοντας αυτό το νομισματικό διάλογο μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση κάνει μια ανάλυση, υπολογίζει τις επενδύσεις που αν είχε ληφθεί η διαφορετική απόφαση της ΕΚΤ, ποια θα ήταν η διαφορά. Και ποια είναι η μεγάλη σημασία της δράσης της ΕΚΤ για την υποστήριξη των ε, επενδύσεων και ότι χωρίς συμβατική και μη συμβατική νοσμοτική πολιτική οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη θα είχαν καταρρεύσει ε, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Βέβαια υπάρχει και η ανάγκη για να προωθήσουμε την πλήρη ανάκαμψη μέσω συνόλου μέτρων που πρέπει να ξεπερνούν τα όρια της νομισματικής πολιτικής, κάτι που θυμίζει πάντα ο Πρόεδρος κ. Ντράγκη. Τέλος, εξίσου σημαντικό, γνωρίζουμε ότι μεθαύριο γίνεται το δημοψήφισμα για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα παραμείνει, θα αποχωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζουμε όλοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσης και η ΕΚΤ είμαστε όλοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οδήποτε αποτέλεσμα και να ε, αντιμετωπίσουμε οδήποτε προβλήματα ε, ισορροπιών. Κύριε Ντράγκη, έχετε το λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που επανερχόμαι στην Επιτροπή σας για την δεύτερη ακρόαση φέτος. Να πω πρώτα απ' όλα πως η ΕΚΤ σημειώνει την σημερινή απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέληξε ότι το πρόγραμμα απευθείας χρηματικών συναλλαγών είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο και εντός της εντολής μας. Στις σημερινέ μου παρατηρήσεις θα εξετάσω την κατάσταση της ανάκαμψης της Ευρωζώνης και τα τελευταία μέτρα νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μετά, κατόπιν ετήματος της Επιτροπής σας, θα συζητήσουμε τις, επενδυτικές προοπτικές αναλύοντας συγκεκριμένα γιατί χρειάζεται περισσότερη δράση για να αυξηθούν οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις, η ανάκαμψη της ε, Ευρωζώνης ε, άρχισε να αποκτά μια ορμή στην αρχή του έτους. Αναμένουμε να συνεχίσει με έναν μέτριο αλλά σταθερό ρυθμό ο οποίος θα στηρίζεται σε στιβαρή εγχώρια ζήτηση και στην ε, αποτελεσματικότητα των μέτρων μας τα οποία θα φανούν στην πραγματική οικονομία. Οι κατανολτές ωφελούνται ακόμα από τις σχετικά χαμηλές ε, τιμές του πετρελαίου και τις βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης. Παρομοίως και οι επενδύσεις αυξάνονται σταδιακά, στηρίζονται από τα υψηλότερα εταιρικά κέρδη και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης. Στο μέλλον, σύμφωνα με τις προβολές του Ιουνίου 2016 του προσωπικού της τραπεζάς μας, το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6% φέτος και 1,7% τα επόμενα δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός ε, στην Ευρωζώνη παραμένει αρκετά χαμηλός. Ήταν ελαφρώς αρνητικός τον Μάιο και αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Ενώ συνεχίζουν οι χαμηλότερες ε, τιμές ε, του πετρελαίου να κρατούν χαμηλά τον πληθωρισμό. Αλλά οι πιέσεις οι εγχώριες, ιδιαίτερα από την αύξηση των μισθών, επίσης παραμένουν χαλαρές, κάτι το οποίο δείχνει μια γενικότερη οικονομική χαλαρότητα. Σύμφωνα με τις προβολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί ε, περίπου στο τέλος του έτους. Κατόπιν αναμένουμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο 1,3% το 2017 και 1,6% το 2018. Καθώς θα ισχυροποιείται η ανάκαμψη και θα κινητοποιηθούν να αδρανής. Από την αρχή των μέτρων χαλάρωσης ε, της ε, πίστης ε, τον Ιούνιο του 2014 τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού έχουν πέσει κατά 80 και 90 μονάδες βάσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιστοίχως και έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά τον Απρίλιο του 2016. Το 2015 είχαμε μια θετική ανάπτυξη της ε, πίστοσης στις ε, επιχειρήσεις της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα Βεβαίως είχαμε και άλλες πηγές οι οποίες ε, ωφελήθηκαν καθώς επίσης ωφελήθηκαν και οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις από βελτιωμένες συνθήκες στις χρηματαγορές, από τα υψηλότερα εταιρικά κέρδη και βεβαίως η χαλάρωση γίνεται ιδιαίτερος αισθητή από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται πολύ σε τραπεζική πίστη στην πρόσφατη μας έρευνα για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση στην Ευρωζώνη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναφέρουν περαιτέρω βελτίωση στην πρόσβασή τους στον δανεισμό και αυξανόμενη προθυμία των τραπεζών να δανείσουν με χαμηλότερα επιτόκια. Τα τραπεζικά δάνεια προς τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις. Επιπλέον θα ακολουθήσει και επιπλέον ε, κίνητρο προς την οικονομία υπό μορφή νομισματικής πολιτικής. Αρχίσαμε επίσης και ένα πρόγραμμα αγοράς ε, στοιχείων από την ε, τράπεζά μας και από την αρχή του 2016 και ειδικά από όταν ξεκινήσαμε και την αγορά εταιρικών ομολόγων τον Μάρτιο οι συνθήκες δανεισμού για εταιρείε με άμεση πρόσβαση στην αγορά ομολόγων έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά. Παραδείγματο χάρη. Το πρώτο εξάμεινο του 2016 το κόστος του χρέους στην αγορά για μη χρηματοπιστωτικές ε, εταιρείες έχει πέσει κατά πέντε μονάδες βάσης. Αναμένουμε και περισσότερες εταιρείες και μέσου μεγέθους να έχουν την δυνατότητα πρόσβαση στην εξωτερική αυτή χρηματοδότηση στο προσεχές μέλλον, καθώς η αγορά εταιρικού χρέους θα επεκτείνεται και θα διευρύνεται. Αύριο θα ξεκινήσουμε την πρώτη λειτουργία μας μιας νέας σειράς ε, μακροπρόθεσμων επιχειρήσεων αναχρηματοδότησης, οι λεγόμενες τέλτρο 2, οι οποίες θα επιτρέψουν στις ε, τράπεζες να έχουν χρηματοδότηση με πολύ ε, ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι θα πλησιάζουν τα επιτόκια τα οποία δίνονται για τις έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα και αυτές με την σειρά τους να βοηθήσουν την οικονομία. Συνολικά τα μέτρα μας έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο να υπάρξει μια στιβαρή ανάκαμψη και να μπορέσει έτσι ο πληθωρισμός να αυξηθεί και να φτάσει σε επίπεδα πιο κοντά στο 2% σε, ένα, σε έναν ε, όχι πολύ μακρινό ορίζοντα. Αυτό φαίνεται επίσης ε, και στην ανάκαμψη της αγοράς διαρκών καταναλωτικών αγαθών που φαίνεται επίσης και στην ανάκαμψη σε επενδύσεις πλήν οικοδομής. Χωρίς λοιπόν τα μέτρα μας αυτά και η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός θα ήταν σαφώς χαμηλότερα. Το πακέτο του Μαρτίου ειδικότερα κατάφερε να αποσοβήσει κινδύνους ύφεση για τις προοπτικέ της Ευρωζώνη. Επιπλέον, όθηση θα δοθεί από τα μέτρα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην φάση της εφαρμογής. Ταυτόχρονα. Η αβεβαιότητα είναι αρκετά υψηλή και οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι ακόμα αρκετά υψηλοί για μια διακοπή της ανάκαμψης λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και της γενικότερης έφραυστης κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της σταθερότητας των τιμών και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας και στην εντολή μας, αν αυτό απαιτηθεί, για να επιτύχουμε τον στόχο μας. Συγκεκριμένα είμαστε έτοιμοι για κάθε εξέλιξη μετά από το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Να πω λίγα λόγια τώρα για τις επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Μετά από τη σημαντική μείωση που παρατηρήθηκε μετά την ε, κρίση του 2008 και την εκ νέου μείωση μετά την κρίση του κρατικού χρέους, οι πραγματικές επενδύσεις στην Ευρωζώνη έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν. Ειδικά οι επενδύσεις των επιχειρήσεων έχουν δείξει μια ανάκαμψη από το 2013 και οι δημόσιες επενδύσεις και οι επενδύσεις σε στέγη έχουν επίσης σε γενικές γραμμές σταθεροποιηθεί. Παρά τις θετικές αυτές τάσεις, ε, το τωρινό επίπεδο επενδύσεων εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό. Το σύνολο των πραγματικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει 10% πιο κάτω από τα επίπεδα προκρίσης, οπότε απαιτείται περαιτέρω δράση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη είναι ένα καλό τέτοιο παράδειγμα. Και θα υποστηρίζαμε την επέκταση του πέρα από το 2018. Η επιτυχία του υφιστάμενου σχεδίου εξαρτάται και από την δυνατότητα να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Και μόνο οι μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα μπορούν να εγγυηθούν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά του στο επίπεδο της Ένωσης. Και εδώ πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει ο συνομοθέτης. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, να εμβαθύνουμε, συγχωρείτε, περαιτέρω την ενιαία αγορά, ιδιαίτερα στην ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιακή οικονομία. Επίσης, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες της υφιστάμενης νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους και συνεπούς εφαρμογής της. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της ρυθμιστικής εφαρμογής θα μειώσει την πολυπλοκότητα, θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού και θα μειώσει και τον κατακαιρματισμό των αγορών προϊόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά έτσι ώστε να διοχετευτούν οι αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις πιο αποτελεσματικά η Τραπεζική Ένωση που περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μάκρο και μικροπροληπτικό ρόλο, έχει ένα σημαντικό ρόλο έτσι ώστε οι τραπεζικές αγορές να κατανέμουν αποτελεσματικά τους πόρους στις πιο αποτελεσματικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρωζώνη. Η πρόοδος στην αγορά των κεφαλαίων επίσης έχει ουσιαστική σημασία για να αναπτύξουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για παραγωγικές επενδύσεις στην Ένωση. Θα βοηθήσει έτσι να βρεθούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης για να τονωθούν οι επενδύσεις ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμα έργα με το να συμπληρώσει την τραπεζική χρηματοδότηση με βαθύτερες πιο ανεπτυγμένες οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν την απλή, διάφανη και τυποποιημένη τιτλοποίηση, αυτά τα οποία δηλαδή συζητάτε τώρα, είναι απτά παραδείγματα του πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να διευρύνει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές εταιρείε να προωθήσει τις διασυνοριακές επενδύσεις και τελικά να έχει θετικό αντίκτυπο στις επενδυτικές προοπτικές της Ένωσης. Στο εθνικό επίπεδο, η μεταρρύθμιση στις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και η μείωση των ρυθμιστικών και διοικητικών στένοπων είναι κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Το συνολικό θεσμικό πλαίσιο μετατρέπει τους ε, χρηματοπιστωτικούς πόρους σε παραγωγικές επενδύσεις που με τη σειρά τους αυξάνουν την παραγωγικότητα και τελικά δημιουργούν δουλειές. Οι αναποτελεσματικές δημόσιες προμήθειες ε, αναποτελεσματικά συστήματα φορολογίας και δικαιοσύνης και το πλαίσιο χρεοκοπίας που έχουν εντοπιστεί σε κάποιες χώρες πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Οι συστάσεις αναχώρα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να βρούμε και να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια σε κάθε χώρα για τις επενδύσεις επιπλέον οι χώρες, ε, τα δημόσια οικονομικά των οποίων το επιτρέπουν, θα πρέπει να προχωρήσουν σε δημόσιες επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη. Για τις λοιπές χώρες να πω πως τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά ωφέλη από πολιτικές που στοχεύουν στην ε, σταθερότητα είναι σοβαρά. τέλο. οι επενδυτές χρειάζονται βεβαιότητα όσον αφορά το οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουν. Αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο πριν από ένα χρόνο σχεδόν, η έκθεση των πέντε Προέδρων παρουσίασε ένα σχέδιο για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Καταλήγοντας, στο μέλλον αναμένουμε να συνεχίσει με έναν μέτριο αλλά σταθερό ρυθμό οικονομική ανάκαμψη. Παρ' όλα αυτά, για να εδραιωθεί αυτή η ανάκαμψη θα πρέπει τώρα οι προσπάθειές μας να εστιαστούν σε ισχυρές δράσεις πολιτικής για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να ευνοηθούν οι επενδύσεις και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Το να έχουμε αποτελέσματα σε αυτούς τους ε, τομείς ε, θα οδηγήσει βεβαίως και τον πληθωρισμό στο να φτάσει σε ένα επίπεδο κάτω αλλά κοντά στο 2% και θα βελτιωθεί έτσι και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων στην Ευρώπη οι πολίτες και οι αγορές πρέπει να είναι σίγουροι για, την δυνατότητες, για τις δυνατότητες μας να ανταποκριθούμε στις κοινέ μας προκλήσεις. Θα πρέπει να εστιάσουμε στο να κάνουμε το κοινό μας σπίτι την Ευρώπη ισχυρότερη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγική σας ε, δήλωση για την πληρέστατη αξιολόγηση των πολιτικών προς αύξηση των επενδύσεων, των επενδυτικών ποσών. Θα δώσουμε το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις. Ο Παύλο Ζάρμα είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δράγκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το Brexit. Είπατε πανελειμμένος πως θα χρησιμοποιήσετε όλα τα πυρομαχικά που έχετε στη διάθεσή σας. Εγώ έχω εμπιστοσύνη γιατί όταν λέτε κάτι το κάνετε στην έκτα. Ελπίζω να μην ε, βγει το σενάριο του Brexit, αλλά ε, παρότι είναι κάτι που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε, αρκεί σε ένα τέτοιο αρνητικό σενάριο μόνο η δράση του ΕΚΤΑ τι άλλο θα έπρεπε να γίνει για να μετριαστεί ο αντίκτυπο μια πιθανή εξόδου τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα για την Καλσρούη και την απόφαση του καστηρίου αυτή η παρακολούθηση ε, εκ μέρους ε, της Γερμανίας του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα επιχειρησιακά ε, τα πράγματα ποια είναι δική σας άποψη και τρίτον ο Μπερνάνκε από τη ΦΕΤ, την Αμερικανική πρόσφατα, είπε ότι υπάρχει μεγάλος ε, φόρτος, μεγάλο βάρος για τις τράπεζες ε, για την ανάκαμψη. Σίγουρα χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και ίσως να μην έχουν όλοι ε, αναλάβει τη δέσμευση που θα έπρεπε να είχαν αναλάβει για τις μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως θα επιθυμούσαμε τουλάχιστον. Εγώ τι θέλω να ρωτήσω, η νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο αν εδώ όλες οι χώρες μέλη είχαν την ίδια δέσμευση και προσήλωση αυτές τις μεταρρυθμίσεις ε, και αν έκαναν όλες οι χώρες τις μεταρρυθμίσεις θα είχε η έκτα περισσότερα περιθώρια ελιγμών σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική. Thank you. Ευχαριστώ. Στην πρώτη ερώτηση να απαντήσω. Δυσχερέστατο να προβλέψει κανείς τις διάφορες διαστάσεις συνεπιών από την ψήφο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πώς θα επηρεαστούν οι οικονομίες και οι αγορές της Ευρωζώνης. Δύσκολο κανείς να κάνει οικασίες ε, ε, για το ποιο αποτέλεσμα θα βγει. Απλώς προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο. Θα ήταν πολύ δύσκολο να είμαι ακριβέστερος τώρα. Κάναμε τη δέουσα προετοιμασία. Για τη δεύτερη ερώτηση. Καταρχάς, το πρόγραμμά μας διατήρησε τη νομισματική πολιτική σε νέο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Λέγαμε ότι πρέπει να εμπίπτει στην εντολή α, ε, της ΕΚΤ η σταθερότητα των τιμών. Κάτι που επιβεβαιώθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σήμερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο στη Γερμανία και το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Τρίτον, μεταρρυθμίσεις και νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική που έχει εφαρμοστεί εξασφαλίζει ότι η κυκλική ανάκαμψη θα λάβει χώρα και λαμβάνει χώρα μάλιστα. Τώρα η κυκλική ανάκαμψη θα μετατραπεί σε διαθροτική. Η απάντηση είναι όχι, χωρίς διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, επανειλημμένα έχω πει ότι έχουμε τη νομισματική πολιτική στα πλαίσια του πληθωρισμού θα επιτρέψει η νομισματική πολιτική να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο στόχο που έχουμε κοντά στο 2%. Η ταχύτητα όμως της επιστροφή σε αυτό το ποσοστό μεταβάλλεται συναρτήση των διαθωτικών αλλαγών. Θα είναι ταχύτερη και λιγότερο δυνηρή διαδικασία αν γίνουν τα δέοντα. Τέτοιες διαθωτικές μεταρρυθμίσεις έγιναν σε κάποιες χώρες. Χρειάζεται όμως περισσότερη δουλειά. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Περβάνος Περέζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, σας ευχαριστώ και για αυτά που είπατε σήμερα και γιατί επιμείνατε στις ε, προκλήσεις ε, και στα πόσα διακυβεύονται στην Ευρώπη, τονίσατε τις επενδύσεις τις Βρυξέλλες είχαμε και το Brussels Economic Forum πριν από λίγες ημέρες και εκεί είπατε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει σαφήνεια ε, και διαφάνεια στην Ευρωζώνη το, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, απαιτείται πρόοδος, ε, μακροπρόθεσμα αλλά και βράχει πρόθεσμα βέβαια λόγω της επίπτωσης ε, για τις επενδύσεις. Αυτά είπατε τότε. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, είστε και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης των πέντε προέδρων, όπου η υπόθεση, το σενάριο για έναν προϋπολισμό της Ευρωζώνης αναφέρεται και όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτησή μας ε, ε, για μια τέτοια πρόταση για, τον για την Ευρωζώνη. Εσείς πώς βλέπετε Ε, αυτό. Τι μέλλον έχει, ανεξαρτήτως της έκβασης του δημοψηφίσματος ε, στη Βρετανία. Επίσης έχουμε την ε, επιμήκυνση του σχεδίου Juncker, του σχεδίου επενδύσεων. Εσείς αναφερθήκατε σε κάποια θέματα. Ε, θα μπορούσαν να εργοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μόνο η έκθεση των πέντε προέδρων, υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν για να ενταχθεί το σχέδιο Juncker σε έναν μηχανισμό. Εσείς μας αναφέρετε ένα παράδειγμα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον θα έπρεπε να γίνουν διορθώσεις ώστε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις δημόσιες επενδύσεις ως ένα είδος μόχλευσης αφενός. Και αν από την άλλη πλευρά θα έπρεπε να επανεξεταστεί ο συντελεστής ε, κινδύνου που προτείνεται, που πιστεύω ότι δυστυχώς ακόμη υπερβολικά προτείνει, ε, προωθεί συγγνώμη, τις επενδύσεις ε, μεγάλης απόδοσης ε, και όχι τόσο αυτές που δεν θα είχαν τόσο μεγάλη απόδοση, αλλά τις οποίες χρειάζεται τόσο πολύ η Ένωση, ιδίω για να υπάρξει σύγκληση των οικονομιών. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Το είπαμε επανειλημμένα. Η Νεοσματική Ένωση εξακολουθεί να είναι ατελής. Και όσο είναι ατελής είναι και εύθραυστη. Εύθραυστη σημαίνει ότι είναι ευάλωτη σε κλονισμούς και τα μέλη, οι πολίτες των μελών αυτής πρέπει να πληρώσουν υψηλότερο τιμήμα για να ανήκουν στην Νομισματική Ένωση από ό,τι θα έπρεπε αν αυτή ήταν ολοκληρωμένη. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η Νομισματική Ένωση. Καταρχάς να είναι πιο ανθεκτική. Να αυξήσουμε την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με άλλο τρόπο. Να αυξήσουμε τον χρηματοστατικό επιμερισμό του κινδύνου. Να ολοκληρώσουμε την Ένωση των Κεφαλαγορών και να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό απορροφής των κλειδονισμών όπως αυτός που υπονοείται στην έκθεση των πέντε πρόεδρων. Καταρχάς, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τις οικονομικές πολιτικές. Είδαμε όταν άρχισε η οικονομική κρίση πόσες χώρες είχαν μια κατάσταση οικονομική, δημοσιονομική που θα τις εμπόδιζε να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε οικονομική πολιτική. Δεν είχαν εργαλεία να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και δεν είχαν τα μέσα να αντιμετωπίσουν την κρίση διότι είχαν ε, καταστήσει πολύ επαχθή την οικονομική πολιτική. η ίδιοι έπραξαν πολλά σφάλματα πολιτικής τα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης. Καταρχάς λοιπόν πρέπει αυτή η οικονομική πολιτική να γίνει ανθεκτική να μην την επιβαρύνουμε υπερβολικά και βέβαια για ασύμε... ασύμετρους κλονισμούς χρειάζεται μηχανισμός απορρόφησης των κλονισμών. Αυτά χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Για να έχουμε δυνατότητα απορρόφηση των κραδασμών χρειάζεται εμπιστοσύνη μεταξύ χωρών. Και για να υπάρχει εμπιστοσύνη, κλίμα εμπιστοσύνη, χρειάζεται αλληλεγγύη μαζί με ευθύνη. Τα δύο πηγαίνουν μαζί. Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο είδη συμπεριφορών Πρώτα απ' όλα τα κάτι μελα συμμορφώνονται με τους κανόνες και δεύτερον θέλουμε τη σύγκληση. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο μέλλον να το συζητήσουμε αυτό, αλλά σας δίνω μια γεύση του πώς το ένα είναι επακόλουθο του άλλου. Πέρα από μια τεχνοκρατική φύσος απάντηση σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Τούτων λεχθέντων. Είναι αυτός ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προχωρήσουμε. Με την πρόσφατη εμπειρία μας μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί ακόμα και χωρίς να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, συναθρήσαμε πόρους για να αντιμετωπίσουμε κοινέ ανάγκες. Παράδειγμα, αντιμετώπιση εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Άλλο παράδειγμα που θα εμφανίζεται όλο και περισσότερο στο μέλλον, αλλά το είδαμε στο παρελθόν, είναι η άμυνα. Διαφορετικός δρόμος αυτός. Αντί να δημιουργούμε θεσμούς και να τους αναθέτουμε καθήκοντα, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενώσεως, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη, αθρίζουν τους πόρους τους για να αντιμετωπίσουν ανάγκες που δημιουργούνται και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που από τη φύση τους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Η δεύτερη ερώτησή σας αφορά τις επενδύσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, αφορά κάτι που είπε επανειλημμένα. Μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις χρειάζονται. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι' αυτό. Τι συνέβη στην κρίση και κάτω από την πίεση των χρηματοστοτικών αγορών. Αρκετές χώρες εξ αυτών ε, προέβησαν σε εξυγίανση δημοσιονομική. Αλλά υπό ακραία πίεση και έτσι διάλεξαν την ευκολότερη δράση τότε. Αύξηση των φόρων έκαναν και περιέκοψαν τις δημόσιες επενδύσεις χωρίς να μειώσουν τις τρέχουσες κρατικές επενδύσεις. Είναι σημαντικό να αποκατασταθούν οι δημόσιες επενδύσεις, το ανέφερα εν είδη εισαγωγής, ότι είναι 10% χαμηλότερο το ποσοστό πριν την κρίση και πριν από την κρίση δεν ήταν ε, υψηλό το επίπεδο, σύμφωνα τα ιστορικά δεδομένα, είχαμε διαδοχικές περικοπές των επενδύσεων δημόσιου τομέα, ξεκινώντα από τα μέσα τη δεκαετία του 90 και μετά. Και αυτό συνέβαινε στις περισσότερε χώρε. Επίσης σημαντικότατο καθίσταται και το εξή. Να είμαστε πολύ επιλεκτικοί όταν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις, να εστιαστούμε στην παιδεία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην έρευνα και το ψηφιακό θεματολόγιο. Περισσότερο αυτά παρά κάποιες απομονωμένες υποδομές. Το σχέδιο Juncker είναι ευπρόσδεκτο. Τα τονίζει αυτά. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η διαδικασία είναι αργή. Δεν παράγει άμεσα αποτελέσματα. Σίγουρα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε την αλλαγή, να αλλάξουμε αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά των προπολογισμών μας, αλλά η διαδικασία είναι αργή και η ΕΚΤ καλωσορίζει και την παράταση πέραν του 2018 της σχετικής διαδικασίας. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, Πίρκο Λέρνερ. Kiitos herra Rahapolitiikan virallisen Σας ευχαριστώ. Φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις μεταξύ των ε, επίσημων ε, πληθωριστικών στόχων ε, των στοιχείων της οικονομίας. Εσείς μας αιτιολογείτε το στόχο για τον πληθωρισμό λέγοντας ότι δημιουργείται οικονομική δραστηριότητα, οι τιμές ε, αν μειωθούν θα επιβαρύνουν την κατάσταση κτλ. Αν ο σχετικός πληθωρισμός είναι πολύ χαμηλός, οι καταναλωτές ε, μειώνουν την κατανάλωση. Η τράπεζα της Φιλανδίας όμως φαίνεται να διαφωνεί Βάσει της ε, Τράπεζας της Φιλανδία ανακάπτει η φιλανδική οικονομία. Λέγοντας, ε, και το υποστηρίζει λέγοντας ότι υπάρχει ε, αλλαγή συμπεριφοράς από τα νοικοκυριά. Υπάρχει περισσότερη ζήτηση, περισσότερη καταναλωτική ζήτηση. Υπάρχουν χαμηλά επιτόκια δανεισμού, λόγω και της δράσης της Κεντρικής Τράπεζας, οπότε έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Μήπως θα έπρεπε να αναθεωρήσετε τους στόχους σας για τον πληθωρισμό, έχοντας υπόψη σας τις προοπτικές της, ρεαλικής, ε, της ε, πραγματικής οικονομίας. Υπάρχει πάντο κίνδυνο υπερβολική δανειοδότηση και δανειοληψία. Αλλά τι κάνουμε με τα νοικοκυριά και πώ εκτιμάτε εσεί τι σημερινέ τάσει. Σα ευχαριστώ. Όπως προείπα, η ανάπτυξη είναι σταθερή, συνεχίζει να υπάρχει ανάπτυξη και η πρόσφατη εμπειρία μας και όχι μόνο μας έχει δείξει ότι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης είναι η αγχώρια ζήτηση κυρίως, άρα η κατανάλωση και οι επενδύσεις ιδίω των επιχειρήσεων που ήταν και βασικός ε, μοχλός ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Αυτά έδειξαν τα στοιχεία μας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής. Και στα μέτρα που λάβαμε από το 2014 ε, τα μέσα του έτους και ίσως ε, και πιο πριν. Επίσης οι τιμές του πετρελαίου βοηθούν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι, όπως σας είπα. Κατά πόσον υπάρχει τώρα ο κίνδυνος περβολικής ε, δανειοδότησης λόγω αυτών των νομισματικών μέτρων. Δεν νομίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε αυτό, όπως σας είπα, το, το φαινόμενο της σταθερής ανάπτυξης τα τελευταία τρία χρόνια. αλλά παρόλα αυτά τα ποσοστά δεν είναι τόσο υψηλά που να δείχνουν ότι θα έχουμε κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης ή υπερβολικής δανειοδότησης. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγης την κατάσταση και την παρακολουθούμε σε συνεχή βάση διότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο δυνατόν νωρίτερα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ramon Tremosa. Ramon Tremosa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό σας μεσημέρι Πρόεδρε Ντράκη, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η εξή. Στην τελευταία σα συνέντευξη τύπου είπατε ότι οι χρηματοοικονομικέ συνθήκε στην Ευρωζώνη ε, είχαν ε, τις, ε, ε, επειδή κάπως δεν ήταν χαλαρές, άλλαξε και η στάση της ΕΚΤ. Είδαμε τα μέτρα του Μαρτίου. Θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές συνθήκες Ευρωζώνης. Δεύτερο, 8 χρόνια από την έναρξη της κρίσης, κάποια κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλό δημόσιο έλλειμμα. Η ΕΚΤΑ πιστεύει ότι οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα με τον ίδιο ακριβώ τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη μόνο στα μικρότερα. Τέλος, τρίτο ερώτημα. Οι πολιτικές της ΕΚΤ σίγουρα βοήθησαν να υπάρξει α, κάποια ανάπτυξη ε, στην πίστη, αλλά δεν βλέπουμε περισσότερε επενδύσει Η ΕΚΤΑ θα στοχεύσουν ε, περισσότερο στο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, να αγοράσουν δηλαδή κάποια ομόλογα ή τέλος πάντων να προωθήσουν τις επενδύσεις ε, δημόσιο ιδιωτικού τομέα. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, οι οικονομικές συνθήκες ήταν αυστηρές, άμα συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Okay. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, οι οικονομικές συνθήκες έγιναν πιο αυστηρές μετά τον Ιανουάριο. Και για μία περίοδο που ήταν πολύ ευμετάβλητη η κατάσταση. Μειώθηκε αυτή η διακύμανση και ανταποκριθήκαμε με το πακέτο που ανακοινώσαμε το Μάρτιο. Αν το δούμε το όλο θέμα με τα σημερινά μάτια, πρέπει τα αποτελέσματα του πακέτου του Μαρτίου να τα αφήσουμε να διαδοθούν, να διαχυθούν στην οικονομία. Εστιαζόμεθα επί της εφαρμογής των μέτρων. Όπως σας προανέφερα, πρέπει να εφαρμοστούν αύριο. Θα γίνει η δεύτερη εφαρμογή τέλτρο και θα εστιαστούμε και επί της αποτελεσματικότητας των προτέρων μέτρων που ενεκρίθησαν. Πώς επηρέασαν την οικονομία τα μέτρα. Χρειάζεται να παρακολουθούμε τις αγορές προσεκτικά. Αν δούμε ανεπιθύμητη ε, συρρήκνωση των οικονομικών συνθήκων, να γίνουν πια αυστηρές οικονομικές συνθήκες, που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τον πληθωρισμό, τότε θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα. Δεύτερο ερώτημα αφορά το έλλειμμα και ότι αρκετές χώρες έχουν υψηλό έλλειμμα. Τι λέγαμε σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς οι κανόνες, με συνέπεια, σε όλες τις χώρες. Έγκαιρα. Η αξιοπιστία των κανόνων είναι θεμελιώδου σημασίας. Θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε αυτό, αν υπάρχουν νομικά ζητήματα που έχουν τεθεί όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, αυτά θα πρέπει να εξεταστούν δεόντως. Το τρίτο ερώτημά σας. Το συζητήσαμε και πριν ίσως. Είδαμε να αυξάνονται οι επενδύσεις. Όπως σας είπα είναι μέτριος ο ρυθμός, αλλά έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ακολουθεί την τάση την ισχυρή για κατανάλωση και επιβιώ... επιβεβαιώθηκε και η τάση των καταναλωτών να αγοράζουν πιο ε, προϊόντα διαρκείας, μακράς διαρκείας. Ευχαριστώ. Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη που παρίσταστε εδώ. Θέλω να επανέλθω στο θέμα των επενδύσεων. Ένα από τα βασικά ζητήματα του διαλόγου είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η επεκτατική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων. Τουλάχιστον όχι στο επίπεδο που θα θέλαμε να δούμε. Διάβασα πολύ προσεκτικά τα διάφορα έγγραφα στα πλαίσια της προετοιμασίας της συνεδριάσεως και ήταν θετική έκπληξη πρέπει να πω λόγω του πλουραλισμού των ε, διάφορων αναλύσεων που μπορούσα να διαβάσω στα κείμενα. Οι ιδέες που βλέπει κανείς στο κείμενο συμφωνούν με τις απόψεις διαφόρων επιχειρήσεων στις διάφορες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και απηχούν οι απόψεις αυτές και τις διάφορες βολιδοσκοπήσεις που έχουν γίνει στις διάφορες εταιρείε. Αλλά οι επικεφαλής των επιχειρήσεων, του επιχειρηματικού κόσμου, αναφέρονται κυρίως στην κατάσταση της οικονομίας και κυρίως στη ζήτηση βασίζονται. Δεν αναφέρονται στη χρηματοδότηση του κόστους ή ε, της πιστώσης και αυτό επηρεάζει τις ε, επενδύσεις. Όταν αναφέρεστε, όταν σας ακούμε να μιλάτε, αισθανόμαστε ότι αυτά που λέτε δεν είναι ακριβώς αυτά που εφαρμόζει η ΕΚΤ. Θέλουμε μια πολιτική που θα τονώσει τη ζήτηση. Θέλουμε κάτι να τονώσει τις επενδύσεις του δημόσιου τομέα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Οι επενδύσεις του δημόσιου τομέα μπορεί να έχουν συνέπειες θετικές και να είναι και θετικά τα πολέσματα και για τα δημόσια ταμεία. Το βλέπει κανείς αυτό σε χώρες όπως είναι η Πορτογαλία. Ακόμα και με τις πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζονται, Ήδη βλέπουμε ότι έχουμε μείωση κατά δύο ποσοστές μονάδες του ελλείμματος σχέση με το 2016, κατά τη διάρκεια του 2016. Ο κ. Δράγκη αναφέρθηκε στην επαναπρόθεση των δημοσίων επενδύσεων. Τα έγγραφα που είδαμε τα πηχούν αυτό. Αλλά οι διεθνωτικές μεταρρυθμίσεις και η πολιτική της ΕΚΤ δεν ταιριάζουν με αυτά που μας λέτε. Σας ρωτώ, έτσι, ευθέως, πώς μπορείτε να ενθαρρύνετε τις δημόσιες επενδύσεις ούτε ότως ώστε να μην χρειάζονται και άλλες διαθετικές μεταρρυθμίσεις. Απάντηση. Καταρχάς, να προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για να σας εξηγήσω ακριβώς ε, πώς έχει η κατάσταση. Εγώ είχα πει ότι ωφελούνται οι καταναλωτές από σχετικά χαμηλές τιμές του πετρελαίου, βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης, επενδύσεις. Επίσης ε, ε, παίρνουν ανωδική πορεία λόγω των κερδών και των, των, συγγνώμη, ευνοϊκών οικονομικών συνθήκων. Για τις επενδύσεις, συγκεκριμένα είπα ότι Είχαμε σημαντική μείωση στη διάρκεια της κρίσης το 2008 και νέα μείωση με την κρίση δημόσιου χρέους στην Ένωση, αλλά οι πραγματικές επενδύσεις στην Ευρωζώνη πλέον αρχίζουν να ανακάμπτουν. Ιδίως οι επιχειρηματικές επενδύσεις που ε, έχουν ευπρόσδετη ανάκαμψη από το 2013 και επίσης δημόσιες επενδύσεις και στον τομέα της στέγασης που μειώνονταν σταθεροποιούνται πλέον. Παρά όμως αυτές τις θετικές ε, τάσεις ε, δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο των επενδύσεων επί του παρόντος γιατί είναι ακόμη κάτω του 10% από τα επίπεδα πριν την κρίση. Αυτά είπα πριν, άρα η νομισματική πολιτική μας αποδίδει υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εφόσον βλέπουμε αύξηση των επενδύσεων. Αυτό αρκεί, όχι δεν αρκεί, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Οι δημόσιε επενδύσεις σίγουρα, α και κάτι άλλο να πω, ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί και γιατί αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. Λοιπόν, να σας πω τώρα, ε, και πριν πω, ε, πριν πω στις δημόσιες επενδύσεις, μιλάμε για την Ευρωζώνη, κατά μέσο όρο. Τι σημαίνει αυτό ότι υπάρχουν ε, περιοχές στην Ευρωζώνη όπου υπολείπονται σημαντικά οι επενδύσεις, ενώ σε, άλλα, ε, σε άλλες περιοχές της Ευρωζώνης οι επενδύσεις ε, πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Οι επενδύσεις. Για να έχουμε επενδύσεις και να πω και κάτι ακόμη, ότι εν γέννη Ούτε και στον υπόλοιπο κόσμο βλέπουμε να είναι πια και σε τόσο καλό επίπεδο. Και σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Και μιλώ τώρα για την Ευρώπη. Χρειάζεται χρόνο γιατί οι πραγματικές ε, αποφάσεις για επενδύσεις χρειάζονται χρόνο. Γιατί υπάρχει και η ανάγκη ενός συγκεκριμένο κλίματος. Δεν πρέπει να υπάρχει αβεβαιότητα, δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια ανασφάλεια. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι επενδύσεις ε, να πάρουν τα πάνω τους. Μας ενθαρρύνει αυτό που βλέπουμε. Αλλά θέλουμε να δούμε ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Σίγουρα οι δημόσιες επενδύσεις έχουν το ρόλο τους και το είπα και πριν. Τώρα, θα μπορούσε οποιαδήποτε χώρα να αποφασίσει να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις. Όχι. Ε, μπορεί να το κάνουν οι χώρες που έχουν δημοσιονομικό χώρο, δημοσιονομικό περιθώριο. Αυτές που δεν το έχουν θα πρέπει να καταρτήσουν τον προπολισμό τους κατά τρόπο ώστε να μειώσουν τις κρατικές δαπάνες και να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις. Και όσο περισσότερο το συζητούμε και ξεκινάμε τα μέτρα, ε, τόσο βλέπουμε ότι η σύνθεση του προπολογισμού είναι πολύ σημαντική. Και το μέγεθος του προπολογισμού βέβαια είναι σημαντικό. Και ιδίως για τις ε, χώρες που έχουν ε, υψηλό χρέος ή μειωμένη πρόσβαση στις αγορές. Για αυτές τις χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουν μια αναδιευθέτηση ε, του προπολογισμού, να αλλάξουν τη σύνθεση του προπολογισμού, ώστε οι δημόσιες επενδύσεις στους τομείς που προανέφερα να αυξηθούν. Πρόεδρος, ευχαριστώ Φίλιπ Λάμπερτς. Καλώς ήρθατε, Πρόεδρε Δράγκη. Τρία ερωτήματα, ELA. Αυτό το προνόμιο των εθνικών κεντρικών τραπεζών που συνάδει και με το γεγονό ότι είναι εθνική και η εποπτεία δεν είναι πλέον όμω εθνική εποπτεία, πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Δεύτερο ερώτημα. Τέλτρο 2. Η πρώτη έκδοση τέλτρο. Υπήρχε ρεσιμότητα που πλέον δεν υπάρχει για την πρόσβαση στο εργαλείο αυτό, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία, αν δεν απατώμε. Ναι, είναι η απάντηση. Υπήρχαν ε, κάποιοι όροι για αυτά τα προγράμματα, ε, στα οποία μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση αν αυξάνει ε, την δανειοδότηση για την πραγματική οικονομία στο τέλκρο 2. Ισχύει αυτό, νομίζω όχι, για πείτε μου για ποιο λόγο. Γιατί ο στόχος είναι να δώσουμε περισσότερη πίστη ε, στην πραγματική οικονομία. Και τώρα έρχομαι στο τρίτο ερώτημα, βασιζόμενο σε κάτι που είπατε και στρέφομαι και στην ε, Περβάς και αυτό που είπε. Είπατε ότι χρειάζεται σύγκληση και συμφωνώ. Αλλά αν πούμε για παράδειγμα μια χώρα όπως είναι η Ιταλία, που την ξέρετε και πολύ καλά. Μετά από 150 χρόνια ε, ενοποίησης δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει και ομοιόμορφη το οικονομικό τοπίο και συνθήκες. Η Γερμανία επανενώθηκε τον ίδιο καιρό με την ε, Ιταλία, 150 χρόνια μετά και με μετά την επανένωση. Είναι τεράστιες οι ανισότητες και οι διαφορές στον οικονομικό ιστό της χώρας. Ναι, συμφωνώ, σύγκληση, καλό πράγμα είναι, αλλά αν το δούμε ε, με την ε, προοπτική του χρονικού ορίζοντα, μπορεί να χρειαστούν αιώνες για να το πετύχουμε αυτό. Η πρώτη ερώτηση για το ELA, η κοινή λογική θα πρότεινε ένα βήμα προς αυτό που υπονοήσατε. Το εξετάζουμε. Δεν είναι απλή απόφαση. Και αυτό διότι είναι ακόμα μια μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις εθνικές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτές είναι αρμοδιότητες που συχνά εφαρμόζονται σε στιγμές ανάγκης και εντάσεων, ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας. Το Διοικητικό Συμβούλιο το εξέτασε αυτό, το συζητούμε, προβληματιζόμεθα επ' αυτού. Δεν έχω όμως κάτι συγκεκριμένο να σας πω περί αυτού ακόμα. Για το τέλτρο 2. Δεν συμφωνώ. Υπάρχει αιρεσιμότητα. Υπάρχει. Το τρίτο σημείο που θίξατε. Είναι σημαντικό τάτο Η σύγκληση λοιπόν είναι θέμα βαθμού συγκλήσεως και σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Όμως η σύγκληση είναι μία από τις βάσεις για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Αυτό που θέλει κανείς είναι να καταβάλλεται συγκεκριμένη προσπάθεια για σύγκληση στην περίπτωση των διαφόρων κρατών μελών, αυτό σημαίνει να αναλυφθούν βασικές μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς. Να καταβληθεί μια ειλικρινής πραγματική προσπάθεια, ούτως ώστε η χώρα και η προσπάθεια της μεταρρύθμισης να φτάσουν στα όρια των βελτίστων πρακτικών. Χρειάζεται χρόνος για κάτι τέτοιο όμως. Δεν το αρνούμε. Τα παραδείγματα που παραθέσατε είναι πολύ καλή απόδειξη ότι χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως, αν αυτή η νομισματική ένωση ε, προβλέπεται να είναι μια ένωση που δεν θα ε, γινόταν μεταφορά. Βασικό θα ήταν η σύγκληση. Εάν δεν υπάρχει σύγκληση, έχεις μόνιμους οφειλέτες και μόνιμους πιστωτές. Η ιδέα είναι να έχουμε ένα στόχο, να έχουμε χώρες που καμιά φορά είναι οφειλέτες, καμιά φορά οι χώρες είναι πιστωτές. Είναι όμως πάρα πάρα πολύ δύσκολος στόχος προς επίτευξη και δεν επιτυγχάνεται σύντομα. Αυτό που θέλει να δει κανείς όμως σε ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα είναι πραγματική αποφασιστική προσπάθεια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάρκο Βαλή Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον Πρόεδρο Ντράγκη για την εισαγωγή του που μας εξήγησε πράγματα σε κάποια σημεία συμφωνούσε για τις δημόσιες επενδύσεις πραγματικά αν καταφέρναμε να επενδύσουμε στην έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία να αλλάξουμε ενεργικέ πηγέ και να δημιουργήσουμε νέες υποδομέ θα ήταν ωραίο. Είδα ότι τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το ΕΦΣΙ, από το Ταμείο Juncker στην Ιταλία, έχουν, ε, αφορούν υποδομή που δεν είναι τόσο βιώσιμη, άρα δεν στηρίζουν την οικονομία. Δύο ερωτήσει έχω. όσον αφορά τον οδικό χάρτη των πέντε Προέδρων, είμαστε στο στάδιο που πρέπει να πετύχουμε συμφωνία όσον αφορά την κοινή εγγύηση για τις καταθέσεις. Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΚΤ σε αυτό το όλο σχήμα των εγγύσεων. Το Federal Reserve μέχρι 250.000 δολάρια εγγυάται στις ΣΥΠΑ για τους τρέχοντες λογαριασμούς η ΕΚΤ δεν μπορεί παρά μόνο μέχρι 100.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί προσπαθούμε να βρούμε ανόητο συμβιβασμό στον αφορά τη στάθμιση του κινδύνου για τα κρατικά ομόλογα όταν θα μπορούσαμε να αντιμαχθούμε εκείνον που θέλει να περάσει αυτό το συμβασμό λέγοντα ότι κάποιε ευρωπαϊκέ τράπεζε έχουν συστημική έκθεση στον κίνδυνο όσον αφορά τα ε, χρεόγραφα, τα αξιόγραφα του τρίτου επίπεδου. Για το βήμα προόδου, το επόμενο ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Πώ πιστεύετε ότι πρέπει να χρηματοδοτείται ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη, Διότι υπάρχουν κάποιε παρουσιάσει, διατριβέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητούμε στην Επιτροπή μα το θέμα αυτό και θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σα. Πώ θα πρέπει να χρηματοδοτείται ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Κατά την άποψή μου, σε μια πραγματική νομισματική ένωση, οι χώρε που απολαμβάνουν το νόμισμα που έχει υποτιμηθεί για την οικονομία, λόγω της οικονομίας και έχουν πλεόνασμα πάνω από αυτό που πετούν οι κανόνες ευρωπαϊκοί, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επανισορροπούν αυτούς τους κλονισμούς κάνοντας μεταφορές πιο σημαντικές έναντι άλλων για να χρηματοδοτούν ε, περιοχές σε ύφεση. Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να λειτουργήσει. Εσείς έχετε αυτή την άποψη ή η άποψή σας είναι διαφορετική από αυτή που σας παρουσίασα. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, λέει ο κ. Ντράγκη, δυστυχώς δεν έχω λόγο διότι ξεπερνά το, την πραγματικό ρόλο του κεντρικού τραπεζίτου είναι κάτι ειδικό που αφορά τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ε, ποιος είναι καλύτερος τρόπος χρηματοδοτήσεως του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι να έχουμε μακροσκοπική θεωρήση των πραγμάτων, δηλαδή ποια θα είναι η οικονομική η πολιτική. Τώρα είναι, ε, ε, αναπτύσσεται, ενώ τα πρώτερα χρόνια δεν ήταν. Άρα υποστηρίζεται η ανάκαμψη. Μπορούν να ληφθούν περαιτέρω δράσεις σε εθνικό επίπεδο, αναθεωρώντας τη σύνθεση των εθνικών προϋπολογισμών, όπως προανέφερα, ή ακόμα και να υπάρξει και ανάπτυξη και αύξηση εκεί που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όσον αφορά το, το μηχανισμό εκεί των καταθέσεων η ΕΚΤ δεν έχει συγκεκριμένο ρόλο και κανόνα. Έχουμε εκδώσει γνωμοδοτήσεις περί του μηχανισμού. Δεν έχουμε όμως συγκεκριμένη άποψη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, το FDIC, όχι η Fed αποφασίζει. Δεν γνωρίζω ακριβώς όμως ποιος είναι ο θεσμικός μηχανισμός ασφαλίσεως των καταθέσεων στις Ηνωμένες τώρα, όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις έχουν αποτελματωθεί, έχουν κολλήσει. Γιατί, διότι από τη μία πλευρά υπάρχει επιθυμία να μειωθεί ο κίνδυνος, να αφαιρεθεί το στοιχείο του κινδύνου από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών κατόπιν αιτήματος να τεθούν όρια του πόσα κρατικά ομόλογα στη θέση τους οι εμπορικές τράπεζες και από την άλλη πλευρά θέλουμε να προχωρήσουμε και να υπάρξει ένας μηχανισμός και να ελέγξουμε κατά πόσο μπορούμε να απομακρύνουμε τον κίνδυνο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας της τραπεζικής μας ενώσεως και είναι σημαντικό να πετύχουμε κάποιο συμβιβασμό ούτως ώστε οι καταθέσει και οι καταθέτες να αντιμετωπίζονται ισότιμα σε όλη την Ευρωζώνη. Έχουμε δημιουργήσει τον εποπτικό φορέα που αντιμετωπίζει τις τράπεζες και τραπεζίτες ισότιμα, δεν κάνουμε το ίδιο όμως για τους καταθέτες. Άρα νομίζω πράγματι υπάρχει σοβαρή ανάγκη να προχωρήσουμε ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ίσοι όροι που επικρατούν για όλους τους καταθέτες στην ε, Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπάρμπαρα Κάπελου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Σύμφωνα με έρευνα της ε, Bundesbank προκύπτει ότι από το πρόγραμμα δανεισμού της Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει μια έλαφρα αύξηση του πληθωρισμού και φαίνεται ότι 2016 έως 2018 ο πληθωρισμός πραγματι θα αυξηθεί κατά 0,1 έως 1% το έτος. Βεβαίως ε, στην πραγματικότητα δεν στέκουν αυτά γιατί τον Μάιο έπεσαν τιμές κατά 0,1%. Το πρόγραμμα σας ε, δανεισμού για 1,74 3 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως ε, έχει πολύ χαμηλές ε, αποδόσεις ε, την προηγούμενη εβδομάδα δημοπρατήθηκαν ομόλογα του Γερμανικού Δημοσίου με απόδοση που ήταν στο δεκαδικό του ψηφίου και εδώ πέρα βλέπουμε πως οι αγορές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντικατοπτρίζονται και στις αποδόσεις των ε, εταιρικών ε, ομολόγων όπου πληρώνουμε τις ε, εταιρείε για να τους δανείσουμε λεφτά. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι με επιστροφή στην αγορά ομολόγων θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε έναν πανικό πωλήσεων και υπάρχει κίνδυνος φούσκας κρατικών ομολόγων και κίνδυνος για την οικονομική σταθερότητα. Κύριε Πρόεδρε, είπατε κάτι ουσιαστικό την προηγούμενη εβδομάδα σε μια ομιλία στις Βρυξέλλες, στην οποία αναφερθήκατε το πόσο σημαντικό είναι να γίνουν διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, για να έρθει να συμφωνεί η νομισματική πολιτική με την οικονομική πολιτική. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Ποια μέτρα προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Ξέρετε πως ε, δεν εφαρμόζονται όλες οι συστάσεις αναχώρα και είναι χαμηλά τα κίνητρα για να εφαρμοστούν. Ποια μέτρα λοιπόν θα προτείνατε συγκεκριμένα. Thank you. Um, first, uh... Σε ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω λίγα λόγια για τις δικές μας πρόβολες ε, του πληθωρισμού. Οι δικές μας οι προβολές ε, λένε ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Μέχρι το τέλος του έτους ο ετήσιος μέσος όρος θα είναι 0,2% αλλά το επόμενο έτος θα αυξηθεί στο 1,3% το 2017 και 1,6% το 2018. Αυτή η προσαρμογή, η άνοδος του πληθωρισμού, ε, συμβαίνει λόγω των μέτρων μας, μέτρων νομισματικής πολιτικής, της αναμενόμενης ανάκαμψης της Ευρωζώνης. Βλέπουμε πως η αύξηση, η ανάπτυξη ε, συνεχίζεται, βελτιώνονται οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και κάποια στιγμή θα έχουμε μια μέτρια ανάκαμψη στους ε, μισθού που υπάρχει σε ορισμένα μέρη της Ευρωζώνης ήδη αλλά δεν έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και επίσης θα υπάρξουν και κάποια αποτελέσματα τα οποία θα φανούν ε, στο τέλος του έτους λόγω των τιμών του πετρελαίου που θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό από το 0 στο 1,3 κατά τη διάρκεια του επομένου έτους. Τώρα, ε, αυτό είναι βασικά ένας μηχανισμός ο οποίος πηγαίνει από την, ε, ανάπτυ... την ανάπτυξη στον πληθωρισμό και παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως όπως όλοι θα συμφωνούσαμε. Όλοι θα θέλαμε μια πολύ πιο γρήγορη ανάκαμψη της ε, ανάπτυξης και του πληθωρισμού αλλά δεν προξενεί και έκπληξη γιατί είχαμε μια τόσο εκτεταμένη και βαθιά ύφεση ώστε θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Και καθώς ε, σταδιακά θα απορροφούμε την ε, χαλαρότητα αυτή θα δούμε πως ε, και ο πληθωρισμός θα ανταποκριθεί. Επίση, σωστά λέτε πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε γενικές γραμμές δεν προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό και οπωσδήποτε οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν περισσότερο. Αν και ε, δεν είμαι εντελώς απεσιόδοξος, κοιτώντας τα τελευταία δυόμιση χρόνια, είχαμε κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε αρκετές χώρες, οπότε δεν ήταν μία περίοδος χωρίς καμία αλλαγή. Και συμφωνούμε πλήρως με την φύση των συστάσεων της Κομισιόν η μόνη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν και να αναλυφθεί η δράση έτσι ώστε να ε, υπάρξει συμμόρφωση με αυτές τις ε, συστάσεις. Σας ευχαριστώ. Μάρκους Φέρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε πάλι εδώ πέρα. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπατε στις 8 Ιουνίου όταν ξεκίνησε η αγορά εταιρικών ομολόγων και να δούμε το κόστος της νομισματικής χαλάρωσης. Ε, Από αυτό επωφελούνται κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν άμεση πρόσβαση στις αγορές ε, κεφαλαίου που ούτως ή άλλως είχαν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και ταυτόχρονα βεβαίως βλέπουμε πως ε, οι τιμές ε, του κινδύνου ενσωματώνονται και στερβλώνουν την τιμή των εταιρικών ομολόγων. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω με βάση αυτά με ποια κριτήρια αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εταιρικά ομόλογα, πώς αξιολογείται τις επιχειρήσεις ε, τα ομόλογα των οποίων αγοράζεται και ποιες, ε, ποιους κινδύνους είστε διατεθειμένοι να εγγράψετε στον ισολογισμό σας. Η στρέβλωση δε αυτή την οποία ανέφερα είναι ένας παράγοντας τον οποίο συνυπολογίζεται και πώς, αντιδράει η πώς αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν αρχίσουν να αραιώνουν τα ομόλογα με το κατάλληλο προφίλ για να αγοράσετε και κάτι άλλο. Την ε, Πέμπτη ε, έχουμε το δημοψήφισμα σε μια μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακοινώθηκε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Βρετανική Κεντρική Τράπεζα έχουν ένα κοινό σχέδιο για την περίπτωση ε, Brexit Αποχώρηση της Βρετανίας για να καθησυχάσουν τις ε, αγορές. Τι υποχρέωση έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δραστηριοποιείται για την Μεγάλη Βρετανία. Um, το πρώτο ερώτημα αφορούσε το πρόγραμμα με τα εταιρικά ομόλογα. Ξέρετε, υπάρχει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου. Οι αγορές δηλαδή εταιρικών ομολόγων φροντίζουμε να συνάδουν με αυτό το πλαίσιο που ισχύει. Επομένως, αγοράζουμε εταιρικά ομόλογα συγκεκριμένης ε, αξίας, συγκεκριμένης αξιολόγησης και επίσης είμαστε και ουδέτεροι ως προς την αγορά σε σχέση με, αυτές τις, ε, με αυτά τα ομόλογα για να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις που θα μπορούσε να ενέχει αυτό το πρόγραμμα. Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε ομαλά και έτσι εξελίσσεται και με αρκετά μεγάλους όγκους ξεκινήσαμε. Τουλάχιστον τώρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο συγκεκριμένο εμπόδιο στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Τώρα, κατά δεύτερον, κατά πόσον αυτό θα ευνοήσει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και όχι τις ΜΜΕ. Όχι. Νομίζω ότι αυτό που παρατηρούμε σε εθνικό επίπεδο είναι ότι μεγάλες επιχειρήσεις η χρηματοδότηση θα αφήσει χώρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες. Και επειδή οι μικρές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τον τραπεζικό δανεισμό σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες, τους μεγάλους ομίλους, βλέπουμε και τα spread ε, για, την, ε, για το δανεισμό ΜΜΕ να, να εξελίσσονται ε, τοτικά και βέβαια αυτό ξεκίνησε πρωτού ξεκινήσουμε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, αλλά συνεχίζεται αυτή η τάση και αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο κόστος του τραπεζικού δανεισμού για τις ΜΜΕ έχει μειωθεί περισσότερο από ότι το κόστος του τραπεζικού δανεισμού για μεγάλες εταιρείες, για μεγάλους ομίλους. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν απλά ενισχύει αυτή την τάση που ήδη την παρατηρούμε, υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχω να σας δώσω κάποια νούμερα Τραπεζικό δανεισμός, ποσοστά για πολύ μικρά δάνεια, παρότι είναι υψηλότερα από τα μεγαλύτερα, το σπρέδι μεταξύ αυτών των δύο συντελεστών έχει πέσει τον Απρίλιο του 159 μονάδες βάσης και η τελευταία έρευνα για την πρόσβαση ε, τον ΜΜΕ σε χρηματοδότηση για τρίτη ε, συνεχή φορά διαπιστώνει βελτίωση και επίσης βλέπει ότι οι τράπεζες είναι πιο πρόθυμες να δανείσουν. Αυτά είναι στοιχεία μέχρι το Μάρτιο του 2016, τα τελευταία μας αποτελέσματα, τα πιο πρόσφατα. Δεύτερο, α όχι, ε, ποιο ήταν το ερώτημα, αν έχουμε κάποιο σχέδιο για να συνεργαστούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε, υπάρχουν εκτεταμένες διαβουλεύσεις ε, μεταξύ όλων των μεγάλων τραπεζών ε, στον κόσμο και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σχέδια όμως, δεσμεύσεις κτλ. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι. Thank you. Σας ευχαριστώ, Χώνας Φερνάντες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πλεόνασμα ε, για τους μας λογαριασμούς αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Είναι ένα πλεόνασμα το οποίο σίγουρα ε, περιπλέκει τα, τους στόχους μας για τον πληθωρισμό. Διότι έχουμε όλες αυτές τις... Ε, ε εκτιμήσεις για το ευρώ. Υπάρχει κάποιο είδους διαχείριση του πλεονάσματος ή του ελλείμματος ε, των διαφόρων κρατών μελών. Δηλαδή, ε, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον θεωρείτε σκόπιμο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου να υπάρχει ένα όχημα με μεγαλύτερη δυνατότητα επηρεασμού για επανεξισορρόπηση αυτών των ε, πλεονασμάτων ή ελλημάτων, κυρίως για βελτίωση των επενδύσεων συνολικά για την Ευρωζώνη το δούνου του τώρα. Έκανε μελέτες αντικτύπου για τα σχέδια διάσωσης σε διάφορες χώρες όπως η Ελλάδα και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η ΕΚΤ θεωρεί σκόπιμο να κάνει και αυτή ανεξάρτητη ανάλυση της δικής της δράσης σε ό,τι αφορά αυτά τα σχέδια διάσωσης. Τέλος, σε μια προηγούμενη απάντησή σας είπατε ότι οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμόζονται on time, είπατε, Εγκαίρω. Αυτό μήπω ήταν ε, μια κρυφή κριτική στη στάση τη Ισπανίας, για παράδειγμα, ή κάποιον άλλον χώρο, δεν ξέρω. Ή αυτό δεν ήταν ο στόχο σα. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Thank you. On your last question, ευχαριστώ για την τελευταία ερώτηση. Θα πω πως οι κανόνες έχουν νόημα αν εφαρμόζονται συνεπώς σε όλες τις χώρες ε, και σε βάθος χρόνου. Και το όφελος των κανόνων υπάρχει ε, αν ενισχύουν την αξιοπιστία του συνολικού ε, χρηματοπιστωτικού πλαισίου, κάτι το οποίο θεωρούμε έναν πυλώνα, θα έλεγα, σταθερότητα για την Ευρωζώνη. Και αν υπάρχουν νομικά θέματα για την εφαρμογή, νομίζω πρέπει να απευθυνθούν εκεί όπου πρέπει. Το είπα και πριν. Τώρα, για μια ανεξάρτητη μελέτη της ελληνικής διάσωσης, ναι, μπορούμε να το δούμε. Δεν έχουμε λάβει κάποια απόφαση, δεν έχουμε συζητήσει κάτι τέτοιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τα μεγάλα πλεονάσματα τρέχουσών συναλλαγών. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ και πολλά χρόνια τέτοια πλεονάσματα και θα έλεγα πως η ιδανική σύνθεση της συνολικής ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια, με χαμηλότερο πλέον τρεξών συναλλαγών και μεγαλύτερη εσωτερική ζήτηση. Για διάφορους λόγους αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά και για τους λόγους που ανέφερα στην εισαγωγική μου δήλωση. Δηλαδή, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, η οποία αποτελεί βάση της ε, ανάκαμψης, ε, μπορεί πράγματι να συμβεί τα επόμενα έτη. Οπότε προβλέπεται ότι με την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης θα μετριαστεί και το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών από μόνο του και βεβαίως το κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων της Ευρωζώνης το οποίο θα ανέβει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Εστέρ Να Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη πολλές φορές ε, μας έχετε πει πως παρά τις μεγάλες συζητήσεις που γίνονται για τα νομισματικά ζητήματα, η νομισματική πολιτική έχει τα όρια της και μιλάτε για την ανάγκη επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για το δεύτερο, μπορείτε να μας πείτε τι είναι πιο επίγον κατά την άποψή σας, ποιες μεταρρυθμίσεις και σε ποιους τομείς για να έχουμε μια πραγματική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, είπατε πως μπορεί να υπάρξει περισσότερη ε, νομισματική να υπάρξει να, υπάρξει ένα πρόγραμμα νομισματικής ε, ενίσχυσης της ε, οικονομίας. Δεν ξέρω. κάποιοι περιμένουν να μπείτε στο ελικόπτερο και να αρχίσετε να μοιράζετε λεφτά. Δεν ξέρω τι πιλότος είστε, αλλά γιατί ακριβώς ε, κίνητρα μιλάτε στην οικονομία και πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τέτοια κίνητρα αν ε, αυτά τα οποία είπατε, δηλαδή ο πυλώνας σταθερότητας που αναφέρατε ή οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αν θέλετε το σημείο που θα προσγειωθεί το ελικόπτερό σας ε, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, οι θετικές μεταρρυθμίσεις η κάθε χώρα έχει το δικό της πρόγραμμα. Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε ποιες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση. Υπάρχουν χώρες που έχουν μία οικονομική δομή που απαιτεί κάποιες αλλαγές για να γίνει ανταγωνιστική και να παραγάγει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και υπάρχουν άλλες χώρες όπου χρειάζονται διαφορετικού τύπου αλλαγές. Κάποιες χώρες χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στο προϊόν, στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Άλλες χώρες χρειάζονται αλλαγές στην αγορά εργασίας. Πολλές χώρες πέραν αυτού χρειάζονται καλύτερη εκπαίδευση, δεν πρέπει να ρωτάμε απλώς γιατί η ανεργία είναι τόσο υψηλή. Μόνο λόγω της ανεπαρκούς ζητήσεως ή αυτό οφείλεται και σε διεθνωτικά αίτια. Αν πάμε στη, στα χρόνια πριν την κρίση, το 2007 περίπου, η ανεργία για την Ευρωζώνη δεν ήταν και τόσο μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα. Πόσο ήταν, 9% νομίζω αν Αυτό δείχνει ότι ίσως δεν είναι μόνο πρόβλημα ζήτησης, αλλά είναι και πρόβλημα δοπο, δομών. Μετά, γιατί η ανεργία των νέων είναι τόσο υψηλή. Αυτή είναι άλλη ερώτηση. Αυτό οφείλεται πιθανότατα σε κάποιες νομοθεσίες σε περί αγοράς ε, εργασίας που αρχές της δεκαετίας, ε, το 2000 περίπου, θεσπίστηκαν και η παιδεία δεν παράγει τα αναγκαία προσόντα. Γιατί τα πραγματικά εμερομίστια ή κάποιες νέες χώρες είναι τόσο χαμηλά. Κάποιες χώρες έχουν πάει στον περασμένο αιώνα, τέλης δεκαετίας του 80. Εκεί οι απαντήσεις θα οδηγούσαν σε έναν κατάλογο αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν. Άλλο κατάλογο. Σε άλλε χώρε είναι πρόβλημα του δικαστικού τομέα. Αν χρειάζονται πολλά χρόνια για να εκδικαστεί μια υπόθεση, όλο το κόστος που αφορά το κράτος δικαίου και την εφαρμογή αυτού θα είναι πολύ ψηλό και θα το πληρώνει η κοινωνία στο σύνολό της το κόστος. Τι λέω, αυτά είναι παραδείγματα των πολλών μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται σε πολλές πολλές χώρες. Για το δεύτερο ερώτημα, με ρωτήσατε αν έχουμε προγραμματίσει και άλλη ε, νομισματική τόνωση ε, που προγραμματίζεται, ανέφερα την Τέλτρο. Τώρα πρέπει να εστιαστούμε επί εφαρμογής, είπα. Βλέποντας τα πράγματα σήμερα, οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και αυτές που θα δρομολογηθούν αρκούν. Αρκούν ούτως ώστε να κατευθύνουν το ποσοστό της ανεργίας κάτω από το 2% αλλά κοντά στο 2% ενδεχομένως να δημιουργηθούν και κατάλληλες προσδοκίες. Αυτό εννοούσα πριν. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέτερ Ζήμων. Κύριε Ντράγκη, πριν σε μία απάντησή σας ε, σε ερώτημα του κυρίου Βάλε τοποθετηθήκατε για την ασφάλιση των καταθέσεων και μας είπατε πόσο σημαντικό είναι να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους και αυτό ακριβώς προσπαθεί η Κομισιόν. Και η επιτυχία βλέπετε πως είναι περιορισμένη. Υπάρχει μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Μήπως θα πρέπει να θέσουμε έναν κοινό στόχο. Δηλαδή ότι θα πρέπει σε όλες τις χώρες το ποσό το οποίο εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι το ίδιο και η εμπιστοσύνη όλων να είναι ξεκάθαρη ακριβώς για αυτό το εγγυημένο ποσό. Και δεν θα έπρεπε ταυτόχρονα ο στόχος να είναι να πούμε ότι όταν ανέβει το η εμπιστοσύνη σε κάποιες χώρες δεν επιτρέπεται παρόλα αυτά να υπάρξει υπαναχώρηση της εμπιστοσύνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας. Αν συμφωνήσουμε, αν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο, τότε ε, αμφιβάλλω αν πρέπει να έχουμε αναγκαστικά τους ίδιους κανόνες για όλους σε όλους ε, τους τομείς. Παραδείγματος χάρη, στην Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν υπόψη τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται σε πολλές χώρες που εμποδίζουν τη χρεοκοπία επιχειρήσεων. Σε πολλά κράτη-μέλη, λοιπόν, υπάρχουν τέτοια μέτρα. Στη Γερμανία έχει ένα όνομα, σε άλλες χώρες διαφορετικό. Ε, μέτρα τα οποία με τη νέα πρόταση δεν θα είναι δυνατά. Ταυτόχρονα όμω προτείνει μέτρα τα οποία λειτουργούν καλά σε ορισμένες χώρε να μεταφερθούν σε άλλες. Πώς θα θέλετε να έχουμε ίδιους κανόνες για όλους αντί να έχουμε έναν κοινό στόχο τον οποίο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε με διαφορετικά μέτρα. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια αποσταθεροποίηση των κρατών μελών εκείνων όπου υπάρχει ε, λιγότερη εμπιστοσύνη των καταθετών. Κοιτάξτε, να σας πω, εν γέννη, και η μείωση του κινδύνου και επιμερισμός του κινδύνου είναι διόψεις του ιδίου νομίσματος και αμοιβαίως ενισχυόμενοι πυλώνες και δεν θα πρέπει ο ένας να είναι προϋπόθεση του άλλου και οι δύο συμβάλλουν στον ίδιο στόχο, δηλαδή ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης. Σημειώθηκε πολύ ικανοποιητική πρόοδος την τελευταία διετία ενισχύοντας Τραπεζική Ένωση με τη δημιουργία του SSM, με την πλήρη αξιολόγηση κλπ. Τώρα, οι περισσότερες τράπεζες Ευρωζώνης πληρούν τα κεφαλου... τις κεφαλουχικές απαιτήσεις. Στόχος τώρα ίσως είναι να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα αναβληθεί επί αόριστον η στόχου. Πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος διαφόρων σταδίων, ένας προγραμματισμός που θα συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία για την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης. Ο κατάλογος θα πρέπει να είναι ορισμένος, να περιορίζεται σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με το ίδις και να μην αναφέρονται σε ε, συζητήσεις που συνεχίζονται με ασαφές χρονικό όριο λήξος. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εφαρμογής του DSG και του BRD και της εναρμονίσεως των διαφόρων άλλων μέτρων και να γίνει και νομοθετική ε, εργασία η κατάλληλη εντός του CRD4. Υπάρχει χρόνος για αυτός, διότι σταδιακή εφαρμογή προς το πλήρες πρόγραμμα της επιτρέπει την πλήρη ε, πρόοδο για να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες για όλους και για να μειωθούν οι κίνδυνοι για τον τραπεζικό τομέα. Τώρα αναφερόμαστε περισσότερο σε μια διαδικασία ποια θα μπορούσε να είναι η μελλοντική διαδικασία τους επόμενους μήνες ούτω ώστε να μην καθυστερούμε επαόριστον. Εκεί πρέπει να δώσουμε προσοχή ενδεχομένως. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ο Γκούναρ Χόκμαρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για την ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης ε, το βασικό, το πρώτο βήμα δεν είναι όλοι να σέβονται τους κανόνες. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα στη Βρετανία. Μας είπατε ότι η ΕΚΤΑ ε, προετοιμάζεται. Για ποιο πράγμα όμως πρέπει να μας πείτε. Αυτό θα ήταν το ενδιαφέρον. Αν αποφασιστεί Brexit, έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας και για τις χρηματαγορές θα υπάρξει μεγάλη ανασφάλεια γενικώ. Και στο City υπάρχουν πολλοί που είναι ισχυροί και στην Ευρώπη που είναι αδύναμοι, αλλά και χρονικά όλο αυτό θα κρατήσει όχι κάποιους μήνες. Μπορεί να έχουμε κάποιες άμεσες αντιδράσεις βραχυπρόθεσμες, αλλά μακροπρόθεσμα θα επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας σε σχέση με τα προβλήματα για τα οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι και ο ΣΑ και το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και άλλοι προβλέπουν μακροπρόθεσμη ύφεση και αυτό σίγουρα θα πλήξει σκληρά τις οικονομίες μας. Τέλος, για την νομισματική πολιτική. Δυσκολεύομαι, οφείλω να σας πω, να, καταλαβα... να καταλάβω γιατί χαμηλότερες ε, τιμές του πετρελαίου ή για την ψυχικη οικονομία ε, μας αναγκάζουν να αυξήσουμε το πληθωρισμό ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ανταγωνιστούμε όταν ε, έχουμε χαμηλούς μισθούς και αυξανόμενη ε, προσφορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχω καταλάβει τη λογική χαμηλή μισθή εκεί, αυξάνουμε εμεί του δικού μα. Ε, δεν έχω καταλάβει πολύ καλά τη λογική και ξέρετε και ποιοι είναι οι λόγοι για αυτέ τι ε, χρηματοπιστωτικέ ε, φούσκε. Η απάντηση για το Brexit. Προείπα ότι δεν θέλω να προδικάσω σε καμία περίπτωση την έκβαση του δημοψηφίσματος. Εμείς παρακολουθούμε ουσιαστικά όλες τις ε, εξελίξεις ε, νομικές, πολιτικές, μεσονομικές και οποιοδήποτε άλλου είδους, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε τις εξελίξεις και είμαστε προετοιμασμένοι για πανενδεχόμενο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα καθημάς, αυτό που θέλουμε είναι να σταθεροποιήσουμε τις αγορές, να παράσχουμε ρευστότητα Έχουμε τις ε, γραμμές ε, σοπ ε, με άλλες τράπεζες και έχουμε και κάποιες διευθετήσεις για τη ρευστότητα που δεν θα δημιουργηθούν τώρα, τις έχουμε. Τις ρυθμίσεις αυτές ήδη σε ισχύ και θέλουμε να χρησιμοποιηθούν με επαρκή τρόπο και να είναι αποτελεσματικές. Είναι σαφές ότι θα προκύψουν και πρόθεσμε και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις με το δημοψήφισμα. Και δεν μπορούμε τώρα ούτε να προδικάσουμε, ούτε να πούμε τι δράση θα αναλάβουμε ανάλογα με τα σενάρια. Λυπούμε για την απάντηση αυτή. Δεν θα τη βρείτε ικανοποιητική ασφαλώς, αλλά έτσι έχει κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το άλλο σα ερώτημα, ουσιαστικά γιατί οι τιμές του πετρελαίου. Ακούστε, στην αρχή όταν οι τιμές του πετρελαίου πρέπει να το έχετε υπόψη το πόσο πέσανε οι τιμές του πετρελαίου ήταν 100 δολάρια το βαρέλι το 2014 και τότε λόγω αλλαγές ε, στην ε, προμήθεια είχαμε πολύ μεγάλη πτώση και αρχές του 2015 και το είχαμε πει και από το 2014 όχι εμείς μόνο όλοι, είχαν πει ότι οι χαμηλές τιμές πετρελαίου είναι κάτι θετικό για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Το 2015 όμως ε, άρχισε και η ζήτηση ε, και όχι μόνο προσφορά να παίζει ρόλο. Οι τιμές δηλαδή άρχισαν να πέφτουν όχι μόνο λόγω τη ε, προσφόρα, αλλά και τη ζήτηση, που ήταν ανεπαρκή. Και αυτό φυσικά είχε να κάνει και με την ανάγκη να στηριχθεί ανάπτυξη στην Ευρωζώνη τέλειο Ιανουαρίου έπιασε το χαμηλότερο επίπεδο 12 ετία στο πετρέλαιο. Έχουμε 80% αναπήδηση στο Brent και έχουμε και το σχιστολιθικό πετρέλαιο στη ΣΥΠΑ. Ε, δεν βλέπουμε και πολύ εξελίξη από εκεί. Υπάρχει υψηλότερη ζήτηση. Υπό την έννοια αυτή, η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου που παράγεται από την υψηλότερη ζήτηση είναι θετικό, θετική εξέλιξη για την Ευρωζώνη. Και με αυτή την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου περιμένουμε, όπως είπα, και ο πληθωρισμός να ε, πιάσει το στόχο μας για το 16, 17 και 18. Άρα, συνολικά, οι εξέλιξεις ήταν θετικές. Τώρα, μια πρόσφατη ανάλυση του Δούνου του δείχνει και επειδή και το Δουνουτού και άλλοι θεσμοί μπορούν να μετρήσουν ε, τον αντικτυπώ στην ανάπτυξη, το ερώτημα είναι γιατί η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου δεν έδωσε τόσο μεγάλη όθηση ώστε να έχουμε την παγκόσμια ανάπτυξη που θα αναμέναμε πριν από κάποια χρόνια. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένη η ανάλυση και είναι πολύπλοκη και πολυσχηδής. Ένας λόγος είναι ότι το παγκόσμιο output, η παραγωγή όλων των πετροπαραγωγών χωρών σήμερα είναι μεγάλη. Μεγάλο το output, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν. Γι' αυτό και έχουμε χαμηλότερες τιμές και για το πετρέλαιο και για τις πρώτες ύλε εν γέννη, που επηρεάζει αυτό βέβαια την παγκόσμια παραγωγή, που είναι μεγαλύτερη από τα προηγουμένω. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ευχαριστώ. Thank you, Andrea Ο Ανδρέα Κοτσολίνο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Επιμένω από ενό θέματο. Η έκθεση λοιπόν τη νομισματικής πολιτική και πώ επηρεάζονται επενδύσει. Δεν συζητάμε την αμφασβήτητη αξία που υπενθυμίσατε και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, όμως φαίνεται ότι δεν παράγει τα επεκτατικά, τα αναπτυξιακά αποτελέσματα για τις επενδύσεις, με περιορισμένη ανάπτυξη διαθεσιμότητας πιστώσεων και είναι πολύ πιο σημαντικό ε, η ζήτηση για πιστώσεις ε, και για επενδύσεις, που είναι πολύ δύναμη. Είπατε ότι είναι δευτερογενέ αποτέλεσμα στην εσωτερική ε, οικονομία και η ζήτηση για τις πιστώσεις. Αυτό χρειάζεται και είναι κάτι που επηρεάζει και το ΑΕΠ. Η παρούσα κατάσταση πόσο απέχει από τις προβλέψεις που για τον αντίκτυπο που έκανε η ΕΚΤ όσον αφορά την ανάπτυξη του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης και να ευθυγραμμιστεί η κατάσταση με τις συνθήκες που θέλουμε πληθωρισμό γύρω στο 2%. Τι σκέφτεστε, πέρα που να λάβουμε υπόψη μόνο το μέσο όρο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, να λάβουμε υπόψη και το πληθωρισμό κάθε κράτους ε, μεμονωμένα. Τέλος, ποιοι είναι οι τομείς, οι μακροτομείς, οι οικονομικοί, οι τομείς που θεωρείτε ότι είναι ομοχλός για να υποστηριχθεί μεσοπρόθεσμα η ανάπτυξη και οι επενδύσεις και για να αναπτυχθούν και οι διάφορες περιφέρειες και να αναπτυχθεί και να αυξηθεί και το επίπεδο της απασχόλησης. Απάντηση. Για την πρώτη ερώτηση, νομίζω ότι μπορώ την απάντησα, αλλά θα μπω σε λεπτομέρειες. Βλέποντας τις επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, τι βλέπουμε, ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις ήταν πολύ μειωμένες στην Ευρωζώνη. Βασικός λόγος βέβαια ήταν η χαμηλή ζήτηση και το χαμηλό ε, επίπεδο των κερδών των επιχειρήσεων. Άρα υπήρχε δυναμικότητα που περίσευε, μεγάλο χρέος των εταιριών, αβεβαιότητα και στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βέβαια ε, είχαμε περιορισμούς όσον αφορά τις πιστώσεις. Για κάποια χρόνια δεν υπήρχε πίστοση διαθέσιμη. Βλέπουμε τώρα μία ανάκαμψη, τη διαπιστώνουμε, στις επιχειρηματικές επενδύσεις ξεκίνησε αρχές του 2013. Το 2015, στο τελευταίο τρίμηνο του 2015, αυτός ήταν ο κινητήρια δύναμη, η βασική της ανάκαμψης. Ποιος είναι ο βασικός λόγος. Σίγουρα η νομισματική μας πολιτική, σίγουρα εν γέννη η ανάκαμψη της ζήτησης, σε κάποιο βαθμό χαμηλότερη, μικρότερη χρέωση των επιχειρήσεων, χαμηλότερο χρέος των επιχειρήσεων και το χαμηλό επιτόκιο. Υπήρχαν όμως και κάποια δεσοτικά εμπόδια που επιβράδυναν και επηρέασαν αρνητικά τα διάφορα επενδυτικά σχέδια. Και το σημαντικότερο από τα αποτελέσματα, το πρώτο αποτέλεσμα, είναι το χαμηλότερο επίπεδο αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Και αυτό εξαρτάται βασικά από το εξής. Οι χώρες, και εδώ πρέπει να το επαναλάβω, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να κάνουν τις διαθωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης ή ε, τις δυνατότητες ε, διαφόρων ε, παραγωγικών νεκρών αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε ε, τις διαθροτικές αλλαγές που απαιτούνται. Το άλλο που θέσατε, εάν έπρεπε να εξετάσουμε τις διάφορους πληθωρισμούς των διαφόρων χωρών. Εδώ μπορώ να απαντήσω όπως θα έπρεπε να είχα απαντήσει σε προηγούμενη ερώτηση. Θα σας πω ότι έχουμε στόχο όσον αφορά τον πληθωρισμό. Ποσοστό πληθωρισμού κάτω από το 2% αλλά κοντά στο 2%. Ο λόγος που έχουμε αυτό το στόχο, διαλέξαμε αυτό το στόχο για τον πληθωρισμό το 2003, είναι οι λόγοι μάλλον ακόμα ισχύουν και σήμερα που διαλέξαμε αυτό τον πληθωρισμό. Δεν υπάρχει πιστικό επιχείρημα αλλαγής ενός στόχου που επελέγει από όλες τις κεντρικές τράπεζες ή τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του υπολείπου κόσμου αρχές της ε, δεκαετίας, αρχές του, του αιώνα, του 2000. Και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο, ότι οι αλλαγές στους στόχους μιας πολιτικής, όταν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος, δεν ενισχύει την αξιοπιστία του θεσμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ντανούτα Χούμπνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία αφορά το ότι πρόσφατα είχαμε διεθνή στοιχεία που δείχνουν πως υπάρχει μία έλλειψη υψηλών ποιοτικών στοιχείων ενεργητικού που μπορούν να γίνουν δεκτά ως, ε, στις συναλλαγές ε, ε, μεταξύ κρατών και που συνήθως βεβαίως εκδίδουν οι κεντρικές τράπεζες ή οι υπερθνικοί οργανισμοί με αξιολόγηση 3α και με αυτόν τον τρόπο αν μετρήσουμε την διεθνή ρευστότητα αυτή έχει πέσει από 60% στο 30% από το 2009 μέχρι σήμερα και Βεβαίως ε, τίθεται το ερώτημα του πώς θα αυξηθούν ακριβώς ε, αυτά τα στοιχεία με υψηλής ποιότητας ε, ιδιωτικά ομόλογα ή ε, ομόλογα κεντρικών τραπεζών. Δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγισή σας για την διεθνή ρευστότητα, γιατί θεωρείτε πως ακριβώ εκεί πέρα οφείλεται η μικρή ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου και της παγκόσμιας ζήτησης. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά ένα άλλο θέμα. Υπάρχει. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα από την Τράπεζα της Αγγλίας, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο τις τελευταίες δέκα Δηλαδή, μια ισχυρή μείωση των φυσικών επιτοκίων τα τελευταία χρόνια έφυσε κατά 5% οπότε η δική μου εντύπωση είναι ότι ο αποπληθωρισμός είναι αυτό το φαινόμενο που ανέφερα είναι παράγοντες που εξουδετερώνουν τις προσπάθειές σας με τη μείωση των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Αυτό το διαρθρωτικό μακροπρόθεσμο παγκόσμιο φαινόμενο το συνυπολογίζεται όταν χαράζεται πολιτική γιατί νομίζω ότι θα επηρεάσει και τις ελλείψεις της νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η έλλειψη τέτοιων ασφαλών στοιχείων είναι οπωσδήποτε ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε, ειδικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και Οπωσδήποτε θα το συζητήσουμε και την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας. Μία υπόθεση η οποία έχει μελετηθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας είναι και αυτή. Ε, τώρα είναι νωρίς να σχολιάσω, αλλά γεγονό είναι πως ε, αντιλαμβανόμαστε αυτή την ανάγκη και θα δούμε ε, θα ε, την αντιμετωπίσουμε. Οπωσδήποτε ισχύει στην ε, Ευρωζώνη όπου βλέπουμε ότι σε καιρούς ε, κινδύνου πραγματικά η απουσία ενός αντικειμένου προς επένδυση χωρίς κινδύνους είναι σοβαρή. Για το άλλο το θέμα που αναφέρατε, πράγματι είχαμε αποκλιμάκωση των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για αυτό, μία από τις οποίες είναι ακριβώς η στασιμότητα που υπάρχει και για την οποία πολλά έχουμε διαβάσει. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η θεωρία για την Ευρωζώνη για έναν λόγο γιατί έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε όσον αφορά την παραγωγικότητα πριν να μπορέσουμε να συγκρίνουμε την κατάστασή μας με τις ΙΠΑ ε, όπου δημιουργήθηκε αυτή η θεωρία. Οπότε για τα πραγματικά επιτόκια στο βαθμό που αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ε, ανάπτυξης ε, και τις συνθήκες δυνητικής ανάπτυξης νομίζω λαμβάνεται υπόψη αυτό στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρτσος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μια ερώτηση για τον κύριο Ντράγκη που έχει σχέση με την ε, κατάσταση στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ε, συνέβαλε και ο ίδιος στη σταθεροποίηση της κατάστασης και η εικόνα σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Όμως η σταθεροποίηση δεν μας φτάνει διότι Αναφέραμε πριν ότι οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10% κάτω από το επίπεδο πριν από την κρίση. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πάνω από 50% πιο κάτω από ό,τι ήταν πριν από την κρίση. Επομένως, θα ήθελα την άποψή του πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, το οποίο είναι πολύ, πολύ μεγάλο, ε, διότι ξέρουμε ότι οι τράπεζες δυσκολεύονται, ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στο 60%. Υπάρχει μια υπερφορολόγηση, δηλαδή όλα είναι δύσκολα. Ε, αλλά ποια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι αν δεν υπάρξει μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, σε 6-12-18 μήνες θα μιλάμε πάλι για την ελληνική κρίση. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην Ελλάδα, όπου σταθεροποιήθηκε η κατάσταση, η οποία πράγματι ήταν άκρος δύσκολη. Οι προηγούμενες δράσεις που συμφωνήθηκαν εφαρμόστηκαν και υπήρξε απόφαση από το διοικητικό του ε, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για τις εκταμιές τα προαπαιτούμενα έχουν ολοκληρωθεί. Σίγουρα χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οδηγήσει και θα συνεχίσουν να οδηγούν σε περαιτέρω σταθεροποίηση της κατάστασης και θα δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Και μαζί με αυτό, μαζί με την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, θα δούμε και μια καλύτερη χρηματοοικονομική κατάσταση γενικότερα. Όπως είπατε και εσείς βέβαια, υπάρχουν ακόμη ε, τροτά σημεία, υπάρχουν αδυναμίες, όπως παραδείγματος χάρη έχουμε ε, τους... Ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες, το αναφέρατε κι εσείς. Εδώ χρειάζεται νομοθεσία που θα δώσει τη δυνατότητα στις τράπεζες να διαχειριστούν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δένα και ουσιαστικά να απαλλαγούν από αυτόν τον παράγοντα που και επιβραδύνει τη ε, πίστη, τη χορήγηση πίστης, αποδυναμώνει τις τράπεζες και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να στηρίξουν επαρκώς τον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το γεγονός ότι η κατάσταση της ρευστότητας για μήνες τώρα ε, χαρακτηρίστηκε από έντονη νεκροή καταθέσεων. Ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την ΕΚΤ που και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Άρα μιλάμε για ένα συνδυασμό. Τώρα η κατάσταση είναι τέτοια που πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί εφόσον εφαρμοστούν οι κατάλληλες πολιτικές, οι ορθές πολιτικές και σε εύθετο χρόνο, σταδιακά θα έλεγα, με την επιστροφή της εμπιστοσύνης ε, θα μπορούσε να υπάρξει και, επαρκής, ε, και σταδιακή άρση των ε, ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων, αλλά αυτό θα συμβάλλει και στην ενίσχυση της οικονομίας και στην παναδημιουργία των συνθήκων για πρόσβαση στις αγορές κάτι που ίσχυε ε, πριν ένα μισή χρόνο. Ευχαριστώ, Ιάκομπ Φόν Βαϊστσέκερ. Ευχαριστώ. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι πιο αργή η ανακάμψή μας είναι το ότι οι ισολογισμοί των τραπεζών αποκαθίστανται πιο αργά στην Ευρωζώνη και ρωτάω άρα μήπως η νομισματική πολιτική σε αυτή τη συγκυρία θα πρέπει να ενισχύει για τον αντίκτυπό της ε, στους ισολογισμούς των ε, τραπεζών ειδικά δεδομένων των αρνητικών ε, επιτοκίων που μπορούν να έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είτε θα είναι ενθαρρύνει τις τράπεζες να δανείσουν περισσότερο ή όσες δεν μπορούν να δανείσουν έχουν άλλο ένα αρνητικό σημείο στον ισολογισμό τους και αναρωτιέμαι τι άποψη έχετε. Ε, ευρύτερα βεβαίω υπάρχει το ζήτημα του ποια περαιτέρω ζητή... βήματα θα πρέπει να κάνουμε στην Τραπεζική Ένωση γιατί παρόλα τα stress τεστ η ανάκαμψη των τραπεζών είναι άνηση στην Ένωση. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την απάντηση που δώσατε στον Πετρεσίμων για την εγγύηση των καταθέσεων. Είπατε πως ε, οποιοδήποτε προαπαιτούμενο για την εγγύηση των καταθέσεων θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη σχέση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Πολύ καλή ιδέα. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε μια ακρόαση σχετικά στην Επιτροπή μας και το Μπρούγκελ έλεγε πως ε, υπήρχε αυτή η σύνδεση σε σχέση με το ότι οι, τράπεζες των, ε, ισολογισμοί των τραπεζών είχαν ακριβώς μεγάλο ποσοστό κρατικών, ε, κρατικού χρέους. Mm. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να... Κοιτάξτε, να σας πω σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάλυση μας όσον αφορά τα αρνητικά επιτόκια και πώς ε, επηρεάζουν τους ισολογισμούς. Το 2015 ήταν το πρώτο πρίες έτος με αρνητικά επιτόκια και τα περιθώρια των επιτοκίων κράτησαν αρκετά καλά το 2015, μάλλον αυξήθηκαν. Είμαι σίγουρος ότι θα, θα επηρεαστούν αρνητικά το 2016. Για ποιους λόγους. Είχαμε επιτάχυνση προκαταβολών και τα ομόλογα με, με σπάγια τιμή που ήταν στα χαρτοφυλάκιο των τραπεζών που έδωσαν κερδοφορία και αντιστάθμισαν τα χαμηλά επιτόκια έχουν εκπνεύσει και τώρα η απόδοση ε, θα είναι πολύ πιο χαμηλή. Άλλος περιοριστικός όρος. Υπάρχουν προβλήματα μεταφοράς, μετακυλήσεως των αρνητικών επιτοκίων στους καταθέτες και σε άλλους πελάτες. Αληθεύει ότι σε άλλες χώρες με πιο αρνητικά επιτόκια από ό,τι στην Ευρωζώνη, η εμπειρία τους δεν ήταν τόσο αρνητική. Υπάρχει και το άλλο. Παρόλο που τα αρνητικά επιτόκια θα μπορούσαν εν ευθέτω χρόνο να στριμώξουν κάπως το ισοζύγιο των τραπεζών, δεν επηρεάζουν τις ροές ε, των πιστώσεων. Μπορούμε να το δούμε και αλλιώς. Δηλαδή να πούμε ότι αύξηση όγκου των δανειοδότησης μπορεί να αντισταθμίσει ε, την αρνητική συνέπεια των ετικών επιτοκίων στα περιθώρια. Προβλέπεται αύξηση των πιστώσεων για το 2016 μεγάλη. Αυτή είναι η πρόβλεψη στις τράπεζες. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε, να είμαστε ρεαλιστές στην προσέγγιση μας. Αληθεύει ότι είδαμε αύξηση πιστώσεως για την οικοκυριά να αυξάνεται κατά 2,2% το τελευταίο 12 μήνο με λήξη το Μάρτιο δανειοδότηση επιχειρήσεων αυξήθηκε μόνο κατά 0,8% και παραμένει αρνητικό σε κάποιες δικαιοδοσίες όπως στην Ολλανδία, στην Ιταλία και στην Ισπανία, σε κάποιες χώρες. Όταν γίνονται έρευνες στις τράπεζες, μας λένε οι τράπεζες ότι πιστεύουν θα αυξηθεί η δανειοδότηση των επιχειρήσεων το 2016 και οι πιστώσει στι επιχειρήσει θα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι πιστώσει Και οι επιχειρήσει τέλκρο θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση των αρνητικών συνεπειών των χαμηλών επιτοκίων. Εν γέννη, ξέρετε γιατί. Διότι το τέρτρο για τις τράπεζες που δανείζουν αυτά τα χρήματα και μπορούν να αποδείξουν έχουν δανείσει περισσότερα σε σχέση με κάποιο όριο θα πληρώσουν το επιτόκιο διευκόλυνση κατάθεσης που είναι αρνητικό. Άρα πληρώνονται ουσιαστικά οι τράπεζες για να δανείσουν. Εν γέννη η αδίποτε βελτίωση των οικονομικών συνθήκων στην Ευρωζώνη θα αποτελεί βελτίωση όσον αφορά τα ισοζύγια των τραπεζών, τα κέρδη των τραπεζών θα επηρεαστούν θετικά διότι οι πιστοτικές απώλειες θα είναι χαμηλότερες το 2015 τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι οι πιστοτικές απώλειες μειώθηκαν και αντιστάθμισαν και με το παραπάνω τον χαμηλό ρυθμό αυξήσεως των περιθωρίων όσον αφορά τους τόκους. Άρα είχαμε μέτρια ε, αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών. Οι τράπεζες οι ίδιες προβλέπουν τις ίδιες ότι μπορεί να συνεχιστούν οι ίδιες τάσεις και το 2016. Αυτό είναι το τοπίο. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως ότι δεν είναι ομοιόμορφη αυτή η εικόνα της πραγματικότητας. Υπάρχουν ε, κάποιοι διάμεσοι που επηρεάζονται περισσότερο από τα αρνητικά επιτόκια και άλλοι λιγότερο. Τράπεζες με μεγάλα αποθέματα α, με κόκκινα δάνεια ή που έχουν χαμηλά spreads όσον αφορά τα στεγαστικά τους δάνεια θα επηρεαστούν από τα αρνητικά επιτόκια περισσότερο διότι ε, υπάρχει μία συνδέεται το επιτόκιο δανειοδότησης με κάποιον ε, ανταγωνιστή και αυτά τα περιθώρια κέρδους μειώνονται με τα αρνητικά επιτόκια. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω για να σας δείξω τι στοιχεία έχουμε, να σας δώσω μία γεύση, μία εικόνα και θα πρέπει να προσέχουμε. Η κατάσταση είναι περίπλοκη γνωρίζουμε τον περίπλοκο χαρακτήρα των διαφόρων διευθετήσεων και όταν αυτός ο μηχανισμός μάλιστα θα κρατήσει επί μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι πολύ περίπλοκος. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η άλλη αφορούσε το ίδις. Ποια ήταν η ερώτηση? Α. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Κύριε Ντράγκη, κύριε Ντράγκη, το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τίθεται όλο και πιο συχνά. Γιατί η ΕΚΤ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα δήθεν ανεξάρτητη νομισματική αρχή, εποπτική αρχή των συστημικών τραπεζών, δανειστής των κρατών μελών της Ένωσης μέσω των προγραμμάτων αγοράς κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και μέλος της Τρόικας υπό, την πολιτική, υπό τον πολιτικό έλεγχο του Eurogroup. Σας έχω θέσει επανειλημμένα το ερώτημα πότε θα φύγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την Τρόικα. Όπως σας υπέδειξε από τον Ιούνιο του 2015 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του επί της υποθέσεως σε 62 του 2014. Μια απόφαση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς και, είναι, και αναφέρθηκε επίσης και σήμερα ή το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλστρούης. Μάλιστα, σε σχετική προφορική ερώτηση που σας έθεσα εδώ στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 23 Ενάτου του 2015 για το πότε η ΕΚΤ θα φύγει επιτέλους από την Τρόικα απαντήσατε ότι η ΕΚΤ δεν θα παραμείνει για πάντα στην Τρόικα. Σας ρωτώ λοιπόν ξανά κύριε Ντράγκη, μήπως ήρθε πλέον η ώρα να αποχωρήσει η ΕΚΤ από την Τρόικα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Το Φεβρουάριο του 2015, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, σε ερώτηση τοποθέτηση που είχα κάνει, μου απαντήσατε ότι η επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών στην Ελλάδα, δηλαδή των S&P και ANFAS, θα γίνει, είχατε πει τότε, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Τελικά η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε ήδη και το ερώτημα είναι ότι το Eurogroup παρά τα αυτά αποφάσισε να μην επιστρέψει τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών και, και της ΕΚΟΥΤΟΥ στην Ελλάδα θα τα κρατήσει ο ESM μέχρι το 2018. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή του Eurogroup ή μήπως θα έπρεπε τα ποσά αυτά να επιστρέψουν στην Ελλάδα ούτω ώστε να αποτελέσουν μέρος των δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη στη χώρα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Να συνοψίσω. Στην αρχή η απόφαση ήταν να συμμετάσχουν τα τρία θεσμικά όργανα στο πρόγραμμα προσαρμογής της Ευρωζώνης. Η απόφαση λήφθη το 2010. Η Νομισματική Ένωση δεν ήταν εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει τα κράτη-μέλη που χάνουν την πρόσβαση στην αγορά. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είδαν ζήτησαν συμβουλευτικό ρόλο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΟΥΝΟΤΟΥ. Αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε για να συναθριστούν οι αρμοδιότητες των τριών θεσμών. Κυρίως όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχε αρμοδιότητες στο τομέα και στο τραπεζικό τομέα και στην βιωσιμότητα του χρέους. Επίσης υπήρχε και καλός λόγος η ΕΚΤ να συμμετέχει ε, σε αυτές τις εργασίες ε, διότι επιτυχή προγράμματα βοηθούν επανόρθωση των διάβλων ε, νομισματικής πολιτικής, αποκαθιστούν τη χρηματοστατική σταθερότητα και προετοιμάζουν το έδαφος για μια επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ ο ρόλος της ΕΚΤ αποφασίστηκε στη δευτερογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Six Pack και του Twin Pack, του Two Pack. Το Two Pack θεσπίζει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο της λειτουργίας, τη, τη λειτουργία της ΕΚΤ βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών και της συνθήκης του ESM. Γιατί το λέω αυτό. Διότι όποια απόφαση λαμβάνεται δεν είμαστε εμείς οι μόνοι που αποφασίζουμε. Η ΕΚΤ ίσως να μην ανήκει για πάντα στην Τρόικα, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα η σωστή στιγμή να αλλάξουμε την μορφή, τη σύσταση της Τρόικα. Και δεν εξαρτάται από εμά η λήψη της δέουσας απόφασης, διότι έχει παγιωθεί, αν θέλετε, ο ρόλος στη δευτερογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το δεύτερο ερώτημά σας, νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε τα κάτι μελη του Eurogroup, όχι εμάς, πώς χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά που αναφέρατε, τα κέρδη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτουσέλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ κάποιες μέρες ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ιταλίας, ο Κάρλο Καλέντα, επετέθη κατά του Προέδρου της Κονσούμπ, το λέω για τους διερμηνείς, Εθνική Επιτροπή για τις εταιρείε και για το χρηματιστήριο κατηγορώντας τον πρόεδρο της Κόνσουμπ ότι έβγαλε από δεδεχόμενα ε, κάποια στοιχεία των διαφόρων προοπτικών. Υπασπίστηκε τον αυτό του και είπε ότι το 2012 αποφασίστηκε ότι συγκεκριμένοι όροι που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των τίτλων προσφέρονται στο κοινό μπορούν να περιέχουν μόνο τις πληροφορίες, τις λεπτομερεί που προβλέπουν τον κανονισμό, πληροφορίες που δεν συμπεριλαμβάνουν τις πιθανότητες που υπάρχουν εξέλιξης. Δεν θα ήταν καλό να ξέρουν πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Δεν πιστεύετε ότι είναι σωστό να γνωρίζουμε πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τοποθετηθεί επί της κοινή προτάσεως των τριών αρχών εποπτείας του χρηματοστικού τομέα της Ευρώπης όσον αφορά τον καθορισμό του εγγράφου που θα δίνει τα βασικά στοιχεία για τον αγοραστή, για τον πελάτη των χρηματοδοτικών αυτών προϊόντων, να ξέρει ο πελάτης ε, ε, συγκεκριμένα στοιχεία. Πότε θα είναι η προθεσμία τελευταία απόφαση και ημερομηνία. Και κάτι άλλο. Αυτέ τις ημέρες η κοινή γνώμη στην Ιταλία ενημερώθηκε και πληροφορήθηκε για αυτά που συνέβησαν στη Λαϊκή Τράπεζα της Βιτσέντσα για τις ε, διάφορες ε, χρηματοδοτήσεις που πέρασαν, ε, αποσιωπήθηκαν από την ΕΚΤ αυτές οι συναλλαγές. Αυτή η δραστηριότητα αυτών των χρηματοδοτήσεων συμβαίνει και σε άλλες τράπεζες ιταλικές, χρηματοδοτικά ιδρύματα δηλαδή. Αυτές οι συναλλαγές που δεν είναι τελείως διαφανείς. Δεν θα είναι ικανοποιητικέ οι απαντήσει, λέει ο κ. Ντράγκη. Στην πρώτη ερώτηση νομίζω ότι θα απαντήσω γραπτό. Ε, είναι σαφέ ότι πρέπει να υπάρχει σαφή ημερομηνία για την απάντηση, αλλά θα σα δώσω απάντηση γραπτό για την ερώτησή σα. Δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω για την υπόλοιπη ερώτησή σα που αφορά την Κόνσουμπ. Και η δεύτερη ερώτηση να τη ρωτήσετε θέστε στη, σε άλλο φορέα στο SSM και όχι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριος Μαυρίδης έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τράγκη την προηγούμενη εβδομάδα uh, εκεί που κάθεστε ήταν ο Λόρδος Χίλ. Ο Λόρδος Χίλ, ο Επίτροπος. Και Αναφερόμενο στην Τραπεζική Ένωση, έκανε ένα σχόλιο το οποίο αφορούσε την σημασία της ε, εμπιστοσύνη ε, και του δίκαιου ανταγωνισμού στις ε, τράπεζες και έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις για αυτά τα θέματα για το θέμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων και ο Γιάκο πριν επίσης δεν είχε χρόνο Πρώτα απ' όλα κάνατε ένα σχόλιο για την ίση μεταχείριση των καταθετών και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Νομίζω το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για το ότι δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ε, ιδιωτικές τράπεζες γιατί πρέπει να βρουν κεφάλαιο από τις καταθέσεις και το να γίνει αυτό σε ένα περιβάλλον χωρίς εγγύηση των καταθέσεων σε ένα μικρό κράτος μέλος κοστίζει πολύ περισσότερο από ότι σε ένα άλλο κράτος μέλος. Οι δύο μου ερωτήσεις λοιπόν είναι οι εξής. Από ό,τι φαίνεται, ο χρονικός ορίζοντας ε, για την πλήρη εφαρμογή της εγγύησης των καταθέσεων είναι το 2024. Θεωρείτε πως ο κίνδυνος αναβολής μέχρι τότε αξίζει περισσότερο από το να πιέσετε ως ανεξάρτητο όργανο για να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο συστημικός κίνδυνος. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξής. Οπωσδήποτε η Τραπεζική Ένωση ήταν ε, ένας συμβιβασμός και με τους τρεις πυλώνες και με τον τρόπο τον οποίο ε, συμφωνήσαμε. Εποπτεία, διάσωση, εγγύηση καταθέσεων. Θεωρητικά θα μπορούσε να έχει γίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Βεβαίω τώρα είναι αργά. Θα μπορούσαμε πρώτα να έχουμε πάει σε εγγύηση καταθέσεων και τελευταία να έχουμε τη διάσωση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Είναι δίκαιο για όλους εμάς που δεχτήκαμε τον συμβιβασμό εγκαίρω να σκεφτόμαστε τώρα την αναβολή ακόμη παραπέρα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, από τη σκοπιά της ε, ΕΚΤ οπωσδήποτε δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης είναι... Περιλαμβάνει πολλές σημαντικές δράσεις, μία από είναι η ολοκλήρωση του συστήματος εγγύησης καταθέσεων ως ένα σημαντικό πυλώνα. Αυτή είναι η απάντηση, λοιπόν, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε έναν συμβιβασμό για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνούσα με το ότι θα μπορούσε να γίνει με οποιαδήποτε σειρά. Γιατί, εάν είναι να έχουμε μία εγγύηση καταθέσεων, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ότι εμείς οι πολίτες, οι τράπεζες πληρώνουμε για την ασφάλιση καταθέσεων άλλων τμήματων της Ευρωζώνης σε τράπεζες που δεν είναι δεν αντιμετωπίζουν εξ άντε κίνδυνο χρεοκοπίας. Οπότε υπ' αυτή τη σκοπιά λογικό είναι να προηγηθεί ο ενιαίος επόπτης ε, της ε, εγγύησης των καταθέσεων. Αλλά βεβαίως αυτό δεν αφαιρεί από το πρώτο το οποίο είπατε, ότι ευκταίο θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβασμό για να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Ευχαριστώ. Για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ναι, τι είπατε ότι οι ιδιωτικέ τράπεζε ε, βρίσκουν κεφάλαιο από τι καταθέσει. Ναι, ναι. Υπήρχε μια τράπεζα, μια τράπεζα ιδιωτική στην περιφέρεια, α πούμε στην Ιταλία ή στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, την Πορτογαλία που αντλεί κεφάλαιο από τι ε, καταθέσει, ε, επειδή έχει υψηλότερο κείμενο πρέπει να ψηλυρώσει υψηλότερα επιτόκια. Αυτό δεν είναι δίκαιο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τράπεζα σε μεγάλο κόσμο. Τι εννοείται ακριβώς ε, ότι βρίσκει κεφάλαιο από τι καταθέσεις, υπό ποια έννοια. Οι καταθέτες βάζουν τα λεφτά τους στην τράπεζα και η τράπεζα του πληρώνει το... Ναι, αλλά αυτό, αυτό είναι καταθέσεις, δεν είναι κεφάλαιο της ε, τράπεζας. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, εννοείται ότι τους πληρώνουν, ε, πρέπει να τους πληρώσουν ε, υψηλότερα επιτόκια, μάλιστα. Λοιπόν, Κοιτάξτε, η εγγύηση των καταθεσεών απευθύνεται κυρίως ε, στους καταθέτες. Και δεν είναι σαφές ότι οι τράπεζες θα πλήρωναν τα ίδια ασφάλιστρα ας, ε, πιθανότατα θα πλέον διαφορετικά λόγω της, ε, των διαφορετικών έγγενων κινδύνων σε διαφορετικά τμήματα της Ευρωζώνης αλλά οπωσδήποτε το, το θέμα πράγματι αφορά τους ε, καταθέτες και αυτή θα ήταν η σωστή κίνηση από μέρους τους. Ευχαριστώ. Yes, we make five minutes break. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών, λέει ο Πρόεδρος.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 Okay. So, dear colleagues... Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντράγκη για την ε, συμμετοχή του στο πλαίσιο του νομισματικού διαλόγου ως προδεκτή της ΕΚΤ και τώρα υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου θα Έχουμε τον επόμενο νομισματικό διάλογο. Συνεδριάζει το Συμβούλιο την Πέμπτη, από ό,τι γνωρίζω, και θα ληφθούν ενδεχομένω αποφάσει που μπορεί να μην μπορείτε να μα αποκαλύψετε εντελώ ε, σήμερα εδώ, αλλά κάποιε ιδέε μπορείτε να μα δώσετε. Να δώσω αμέσω το λόγο σε εσά για την εισαγωγική σας παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή Νομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, χαίρομαι πολύ που μπορώ να σα μιλήσω σήμερα από την ιδιότητά μου ω Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Καταρχά, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Γενικό Συμβούλιο του ε, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου θα συνεδριάσει όπως είπατε και εσείς την Πέμπτη και με τα χαρά θα σας ενημερώσω στην επόμενη ακρόαση εδώ για το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων. Ωστόσο θα ήθελα να τονίσω ορισμένες από τις προτεραιότητές μας, ιδίως ε, ε, για κάποιους τομείς τον οποίο νομίζω ότι μπορούμε μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας. Το πρώτο θέμα λοιπόν αφορά τον ε, μεσοπρόθεσμο αντίκτυπο του χαμηλού επίπεδου επιτοκίων αλλά από μάκρο εποπτική οπτική γωνία. Όταν συνεδριάσαμε για τελευταία φορά είχα αναφερθεί ε, στις ε, στο έργο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για τις μεσοπρόθεσμης επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα των χαμηλών επιπέδων των επιτοκίων. Αυτό το εξετάζουμε υπό το διαρθρωτικό πρίσμα, για να δούμε δηλαδή κατά πόσον ε, και με ποιο τρόπο θα επηρεαστούν τα επιχειρηματικά μοντέλα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τραπεζών, ε, ασφαλιστικών εταιριών, συνταξιδοτικών ταμείων, επενδυτικών ταμείων, όπω και υποδομέ αγορά. Φυσικά εξετάζουμε μεταξύ άλλων ε, και την αλληλεξάρτηση με κυκλικούς παράγοντες όπως είναι τα επίπεδα αποδοτικότητας, ε, κερδοφορίας και την ανάγκη εξασφάλισης ε, βιώσιμης απασχολ... Ε, χρηματοδότησης. Συγγνώμη. Το έργο μας εστιάζει πρώτον στον αντίκτυπο του χαμηλού επίπεδου των επιτοκίων στην οικονομία και στη συμπεριφορά των οικονομικών φορέων. Δεύτερον, εστιάζουμε στον αντίκτυπο στις τράπεζες, ασφαλιστές, χρηματοπιστωτικές αγορές και τρίτον στην αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των ε, τομέων. Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που σχετίζονται με τα χαμηλά επιτόκια θα μπορούσαν να αποκρισταλωθούν ε, σε διάφορα ε, σκέλη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, άρα πρέπει να υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση για την χάραξη πολιτικών και προς τούτο εξετάζουμε τρεις βασικές ομάδες κινδύνων. Πρώτον, τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων. Δεύτερον, ευρύ ανάληψη κινδύνων. Και τρίτον, αλλαγές στη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι πολιτικές για την, τον, αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων των δύο κατηγοριών έχουν ως στόχο τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίσεων και την ε, ομαλή έξοδο ε, των θεσμών εκείνων που έχουν μη βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Σε ό,τι αφορά την τρίτη κατηγορία, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι αλλαγές ε, στη δομή ε, της αγοράς μπορεί να αλλοιώσουν τη φύση των κινδύνων και επομένως να χρειαστεί να ορίσουμε μακροπροληπτικές ε, πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Το Γενικό Συμβούλιο του ECRB θα συνεχίσει να συζητά αυτά τα ζητήματα και θα επικυρώσει το τεχνικό έργο αυτήν την εβδομάδα. Όπως είπα, χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για την, ε, σε επιπτώσεις που έχουν ε, τα χαμηλά επιτόκια. Ευρύτερα Τίνια, πιστεύουμε ότι αυτή η ολιστική έποψη είναι ανάγκη και για τη μακροπροληπτική πολιτική την πολιτική της μακροπροληπτικής εποπτείας. Και έρχομαι σε ένα άλλο σημαντικό για το ECRB ζήτημα που είναι η ε, χάραξη μιας στρατηγικής για τη μακροπροληπτική πολιτική πέραν του τραπεζικού τομέα ήδη εφαρμόζεται για τον τραπεζικό τομέα με μακροπολιτική πολιτική, ωστόσο η στρατηγική, τα αριθμιστικά δεδομένα και εργαλεία για την αντιμετώπιση κινδύνων πέραν του τραπεζικού τομέα χρήζουν περαιτέρω βελτίωση, είναι σαφές. Και αυτό είναι ένα καθήκον για το οποίο θα απαιτηθεί συνεργασία μεταξύ ενός ευρέως φάσματος διαφερμένων φορέων. Νομοθέτες, η SRB, μακρο-μικρο-προληπτικές ε, αρχές και ρυθμιστές, ρυθμιστικές αρχές. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι ένα πλαίσιο ανάλυσης και πολιτικής ε, για τη στόχευση των κινδύνων σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα με μία δέσμη μέτρων που μπορεί, πρέπει να είναι μεν συνεπή, αλλά δεν χρειά, μέτρα που δεν χρειάζεται να είναι συνεπή, μάλλον απαραίτητα ομοιόφαλα, αλλά πρέπει να είναι συνεπή, ιδίω μεταξύ άλλων για ασφάλεια με μεταπιστωτικέ αγορές και υποδομή των αγορών. Επίση θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε τομεί με μεγαλύτερο κίνδυνο ε, συστημικό. Επομένως, το απαιτούμενο επίπεδο αντε, αντοχής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ιδίως ε, στα επενδυτικά ταμεία και άλλους τέτοιους ε, τομείς θα πρέπει να συνδέεται με, τη, με τον αντίκτυπο που θα είχαν σε σχέση με τους συστημικούς κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει συνολικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το υπερβολικό χρέος ε, των οικονομικών φορέων. Επομένως, η κίνδυνοι στο επίπεδο των τελικών δανειοληπτών, ανεξαρτήτως του είδους ε, πίστοσης, τραπεζικά δάνεια, μη τραπεζικά δάνεια ή εμπορεύσιμα χρεόγραφα κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ίσως χρειαστεί ανάπτυξη ενός πλαισίου για τις απαιτήσεις μόχλευσης για τα επενδυτικά ταμεία. Καθώς επίσης θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες πηγές δεδομένων που ε, είναι διαθέσιμες ε, υπό την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον προτείνουμε την ανάπτυξη μιας ευρύτερης εργαλειοθήκης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που θα περιλαμβάνει δοκιμές αντοχής top-down για τους διαχειριστές ε, περιουσίας, ε, για τα συνταξιδοτικά ταμεία, τις ασφάλειες, ε, τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και καθώς και για τα πλαίσια εξυγίανσης ε, τη διάσωση για του κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και του ασφαλιστέ. Θα δημοσιεύσουμε σύντομα ένα έγγραφο στρατηγική που ελπίζουμε να είναι σημείο αναφορά για τη χάραξη τη μελλοντική πολιτική. Επιτρέψτε μου τώρα να πω δύο λόγια για τη ρευστότητα και συγκεκριμένα για την αξιολόγηση των κινδύνων σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά ταμεία ε, και, τον, ε, και το λεγόμενο market making sector και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι υπεύθυνοι πολιτικοί αναφέρουν το κατά πόσον, το, θέτουν το ζήτημα το κατά πόσον οι συστημικοί όροι για τη ρευστότητα επιδίνωσαν την κατάσταση και αν έχει κάποιες παρενέργειες ε, ανεπιθύμητες ε, η νέα νομοθεσία. Δηλαδή, απαιτείται πολιτική ε, απάντηση σε ανισορροπίες μεταξύ ζήτηση και προσφορά ρευστότητα, αν υπάρχουν αυτέ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό προληπτικό ζήτημα, γιατί θα μπορούσαν αυτέ οι ανισορροπίε να διευρυνθούν και να μεταφέρουν του κραδασμού σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εμεί επεξεργαζόμαστε την αξιολόγηση κινδύνων σε αυτού του δύο τομείς που σα προανέφερα, investment fund, market making και έχουμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ικανότητα συλλογής δεδομένων ε, και αναλύσεων ε, και ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε συλλέξει 200, στοιχεία για 274 εταιρείε διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, 1668 επενδυτικά ταμεία σταθερού εισοδήματος. Η πρώτη τεχνική αξιολόγηση που βασίζεται στους υπολογισμούς μας μας οδηγεί στο συμπέρασμα το 95% του κλάδου θα μπορούσε σε ένα ακραίο αλλά πιθανό σενάριο να εξαργυρώσει πλήρω αξιώσει. Αυτό το λέω, πρέπει βέβαια να το επιβεβαιώσει το Γενικό Συμβούλιο. Και τώρα σε ό,τι αφορά τις ε, πρόσφατες ρυθμιστικές ε, αλλαγές και το κατά πόσον χωρίς να το θέλουν μπορεί να περάσουν ε, την ρευστότητα στις αγορές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των νέων κανόνων. Δηλαδή, τι σημαίνει ε, αυστηρότερη ρύθμιση σημαίνει ότι μπορεί να απορροφηθούν καλύτερα οι απώλειες όταν η αγορά αντιμετωπίζει πιέσεις, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη αθεκτικότητα, μείωση των ε, αναταράξεων στις αγορές. Ε, σας έχω λοιπόν ενημερώσει τώρα για τις βασικές μας προτεραιότητες και τώρα θα ήθελα να στραφώ ε, σε κάποιες από τις δημοσιεύσεις μας, τις πιο πρόσφατες. Σε ό,τι αφορά το στόχο της ε, ανάπτυξης ενός μακροπροληπτικού πλαισίου για τον τραπεζικό τομέα, πρόσφατα θεσπίσαμε το πλαίσιο για την εθελοντική διασυνοριακή αμοιβαιότητα μακροπροληπτικών μέτρων. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται ήδη για το Βέλγιο και Εστονία πρόσφατα. Επίσης, στην Επιτροπή σας έχω προαναφέρει ότι εργαζόμαστε σε ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε σχέση με τα ακίνητα, εμπορικά και μη. Έχουμε εκθέσεις που δημοσιεύονται. Είναι πλέον, έχουν αναρτηθεί και παρέχουν ένα μοναδικό σετ δεδομένων για τις διαρθρωτικές διαφορές. Επίσης έχουμε δημοσιεύσει μια αξιολόγηση των μακροπροληπτικών πολιτικών σε σχέση με τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες της Ένωσης το 2015 και προτιθέμεθα να κάνουμε το ίδιο κάθε χρόνο. Επίσης, εργαζόμαστε σε σχέση με τις ασφάλειες και είχαμε πρόσφατα την έκδοση μιας έκθεσης του SRB για τους συστημικούς κινδύνους στον τομέα των ασφαλείων στοιχίζουμε το έργο μας για τις ασφάλειες στο ESRB, διότι παρά το ότι συχνά υποστηρίζεται, υπάρχουν συστημικές πτυχές στις ασφάλειες που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Τέλος, η έκθεση της ε, Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής ε, που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο συνεισέφερε σημαντικά στη συζήτηση για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους κινδύνους που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος. Θα θυμάστε ίσως ότι αυτή η έκθεση ήταν ως απάντηση στις ερωτήσεις που μας θέσατε στην Επιτροπή αυτή και σας ευχαριστώ για το θέμα αυτό που δεν γύρατε και να σας, διασφαλ... να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε τους κινδύνους της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που προέρχονται από την αλληλή του κλίματος να τους εξετάσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Σας διαβεβαιώ επίσης ε, ότι θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά και τα ερωτήματά σας για ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που σχετίζονται με την ε, εισαγωγή των ε, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, η FRS 9. Ο Χαβιέρ Σουάρες, ε, προηγείται, ε, ηγείται συγγνώμη, μιας νέας ομάδας εργασίας που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό και θα συνεδράσει για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ε, θετικές πληροφορίες για το διάλογο με το Κοινοβούλιο για διάφορα θέματα και για αυτό που είπατε για την ομάδα εργασίας για το IFRS 9 λόγω χρονικών περιορισμών θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο ερωτήσεων για 1,5 λεπτό και παρακαλώ όλο η ερώτηση και απάντηση να περιοριστεί στα 4 λεπτά. Ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες είναι ο πρώτος που υποβάλλει ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο Μάριο Ντράγκη. Η ερώτησή μου αφορά την Δημόσια Τράπεζα Πορτογαλίας, την CGT, τη μεγαλύτερη Δημόσια Τράπεζα Πορτογαλίας. Η ΕΚΤ έδωσε οδηγίες, ζήτησε από την πορτογαλική κυβέρνηση να αφαιρέσει τα όρια τα μισθολογικά ή να αυξήσει τα μέγιστα όρια των πληρωμών, των μισθών, των διευθυντών της Cash General de Deposito, CGT, και πώς θα διαθέσετε τέσσερα δις ευρώ των φορολογουμένων στην ε, τράπεζα αυτή συνοδεύεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη CGD που ετοιμάζει η τράπεζα ε, ε, το υποστηρίζεται αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί η εδαφική κάλυψη που έχει η τράπεζα ή θα μειωθεί το προσωπικό της τράπεζας, να τα χρήματα. Απάντηση. Καλύτερα να απαντηθεί από την SSM η τράπεζα και όχι από την δική μας ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συστημικού Κινδύνου. Δεν το συζητήσαμε ποτέ. Η κυρία Περβόμος Περέζης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφερθήκατε σε προηγούμενη ακρόαση στο εξής. Για να μπορεί να λειτουργεί το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου καλά, θα πρέπει ε, να ακολουθήσει σωστή προσέγγιση. Σήμερα ε, βασκόμαστε ενώπιον του Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων βρίσκεται ο φορέας σας. Λαμβάνοντα υπόψη τις συνθήκες για τη θέση ισχύ των διεθνών προδιαγραφών, δεν πιστεύετε ότι είναι σημαντικό εν αναμονή της προσαρμογής που γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εργασιών που κάνει η Επιτροπή για τη λειτουργία των αγορών και τη σταθερότητα να μπορεί να τεθεί σε ισχύ το μέτρο το ταχύτερο δυνατόν βάσει της ε, προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, να πω καταρχήν ότι υποστηρίζω πλήρως το καθεστώς διάσωσης των ταπεζών και το βασικό στοιχείο, δηλαδή το bail-in. Ο ενιαίος μηχανισμός διάσωσης είναι συμπλήρωμα της κοινή εποπτείας που έχει δημιουργηθεί και σημειώσαμε θεματική ε, πρόοδο ρυθμιστικά. Όμως ε, παραμένουν κάποια προβλήματα. Το πρώτο είναι αυτό που αναφέρατε, δηλαδή σαφές νομικό πλαίσιο όσον αφορά την απορρόφηση ε, του δυναμικού για τις τράπεζες, το ΜΡΕΛ δηλαδή με άλλα λόγια, και πώς εφαρμόζεται με συνέπεια αυτό το μέτρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κάτι κρισίμου σημασίας. Μετά, ευθυγράμμιση του ΜΡΕΛ με, με το ΤΙΛΑΚ, που είναι το αντίστοιχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα έλεγα λοιπόν ότι εν γέννη το, το Συμβούλιο για τη ε, διαχείριση, ε, για τη διάσταση των τραπεζών είναι πιο καλά εξοπλισμένο. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο που έχει εφαρμογή του ΜΡΕΛ. Πρώτα απ' όλα είναι η σχέση του ΤΙΛΑΚ με το ΜΡΕΛ όσον αφορά τη λειτουργία εφιστόμενων πολιτικών δηλαδή ε, αυτό το σύστημα απορρόφησης των ε, κεφαλαίων μετά ίσως να υπάρχει κίνδυνος διάδοσης κινδύνων και νέοι διάβλη ε, διασύνδεσης στο σύστημα λόγω διαφόρων ευθυνών που λαμβάνονται στα πλαίσια του Μπέιλιν. Μετά, κυκλικές συνέπειες των, της χρήσης του Μπέιλιν Τέταρτον, πρέπει να δούμε πώς είναι οι υποχρεώσεις χρηματοδότησης, οι απαιτήσει έκδοσης ΜΡΕΛ, δηλαδή επιλεξίμων αυτών χρεαγραφών, επηρεάζουν την οικονομική ανάκαμψη και χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Αυτή είναι σφαιρικά λοιπόν η εικόνα των τομέων όπου εκεί θα εκφραστεί το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Ευχαριστώ. Η Κέι Σουίνμπερν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά εκπροσωπή τη Άντρα Λούντς. Την αντιπροσωπεύω, δεν μπορεί να παρίσταται. Θα ζητήσω ερωτήσεις τύπου Ευρωζώνη που δεν γνωρίζω πολύ καλά. Έγινε ε, ε, ε, στο Μάιο του 2016 εξετάστηκαν διάφορα στοιχεία σταθερότητα στην Ευρωζώνη με, με, συστημικό κίνδυνο μέσου επίπεδου βλέπουμε χαμηλό κέρδος, προπτικές κερδών για ασφαλιστές και τράπεζες με τους μεσάζοντες των τραπεζών να περιορίζονται και υπάρχουν προβλήματα ανεπίλητα για τα κόκκινα δάνεια. Φαίνεται ο συστημικός κίνδυνος τελικά έχει τονιστεί περισσότερο σε σχέση με τον προηγούμενο προηγούμενα θεώρηση. Η ΕΚΤ βλέπει αν η πολιτική των κεντρικών τραπεζών εισάγει συστημικό κίνδυνο στο χρηματοστικό τομέα κυρίως στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, η έκθεση εξετάζει τον κίνδυνο που δημιουργείται από τα ανεπίλητα προβλήματα για την μείωση των κόκκινων δανείων. Έχει δημιουργήσει task force η ΕΚΤ για τα κόκκινα δάνεια. Η SRB, το, σύστημα, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, κάνει κάτι πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Το, η μείωση των κερδών των τραπεζών και των ασφαλιστών είναι ένας κίνδυνος βασικός κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. κυρίως στο περιβάλλον των πολύ χαμηλών επιτοκίων. Στην αρχή του έτους παρατηρήσαμε μεγάλες μεταβολές όσον αφορά τις τιμές των χρεογράφων των τραπεζών και είχαμε και χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών λόγω αυτού εν μέρη οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πιέσεις κερδοφορίας λόγω μειώσεως ε, των ε, περιθωρίων των τόκων, το ανέφερα στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες, όπως η ανάπτυξη του όγκου των δανείων, τα εισοδήματα τα τέλη από τις φορές που καταβάσει τράπεζες, τις κρατήσεις τραπεζών και σε κάποιες χώρες το χαμηλό επίπεδο κόκκινων δανείων. Και όσο προχωράει η ανάκαμψη θα περίμενε κανείς υψηλότερη ποιότητα των πιστώσεων, άρα βελτίωση και για, τις, για τα αναπομένοντα κόκκινα δάνεια, αλλά και για την ποιότητα των νέων δανείων. Άρα θα έχουμε αύξηση αποδοτικότητας και μείωση του κόστους. Οι ασφαλιστές τα κατάφεραν καλύτερα από τις τράπεζες, αλλά αντιμετωπίζουν και αυτοί ε, λιγότερα κέρδη λόγω των ε, χαμηλών επιτοκίων. Άρα αναλύουμε όλες τις ε, εξελίξεις και πιο συγκεκριμένα σχεδιάσαμε μια συζήτηση αυτή την πέμπτη όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Συνεργαζόμαστε και με την EBA για το θέμα αυτό, Τάπεζα Ένωση Τραπεζών. Θα, ενημερώνουμε την, ε, θα ενημερώσουμε δεόντως την Επιτροπή σας λοιπόν, ίσως στην επόμενη συνάντηση. Ο Μικαήλ Τόερερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη. Αναφερθήκατε μόλις ε, στο θέμα των ε, χαμηλών επιτοκίων, όχι από τη σκοπιά της νομισματικής πολιτικής, αλλά από τη σκοπιά των μακροδυνητικών κινδύνων. Θα ήθελα τώρα να αναφερθούμε στο ότι δεν είναι μόνο τα βραχυπρόθεσμα αλλά και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια χαμηλά. Και βεβαίω αυτό δεν μπορούν να το επηρεάσουν οι Ευρωπαϊκές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί ε, δεν αφορά καν την ε, Ευρωζώνη. Το ίδιο ισχύει και στην ε, Δανία και στην Ελβετία. Μήπως αυτό οδηγεί στο ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδοτικά επενδυτικά έργα και προϊόντα και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφάλειες ε, ζωής βρίσκονται σε μια φάση χαμηλών τόκων ε, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και το θέμα είναι πως, επίσης η άλλη ερώτηση είναι πως ε, αξιολογείται την κατάσταση του ιδιωτικού χρέους σε σχέση με την οικονομική σταθερότητα. Ευχαριστώ. Να πω πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα. Είπα, είχαν μηδενικά επιτόκια για πόσο, 8-9 χρόνια δεν θυμάμαι. Και κι όμως ο αντίκτυπος ε, στις ε, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείε δεν είναι συγκρίσιμος με αυτό το οποίο ακούμε ότι θα ήταν ο αντίκτυπος ε, στην Ευρωζώνη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, πιθανώς, αλλά και το ότι υπάρχουν κάποιες ρυθμιστικές διατάξεις που επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες ε, να κάνουν διαφορετικές επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις ή ε, οφείλεται στη μεγαλύτερη ευελιξία των επιχειρηματικών μοντέλων κάποιων τέτοιων εταιρείων. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποιος λόγος για αυτά τα χαμηλά επιτόκια. Δηλαδή υπάρχουν για να προωθήσουν την ανάκαμψη και να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Εύρωστη ανάπτυξη και οπωσδήποτε αυτά θα ωφελήσουν τον ισολογισμό τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρείων και ταμείων. Οπότε τα χαμηλά επιτόκια είναι ένα σύμπτωμα το οποίο εμφανίζεται λόγω των γενικών συνθήκων της οικονομίας και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε να προσαρμοστούν στο βαθμό του δυνατού τα επιχειρηματικά μοντέλα. Αλλά γνωρίζουμε πως είναι βεβαίως και ένας παράγοντας ε, κινδύνων ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και το γνωρίζουμε αυτό και στην Κεντρική Τράπεζα και στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις ε, τις σχετικές. Τώρα, να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Αν κρατήσει αυτή η κατάσταση πολύ καιρό, που θα αναζητήσουμε ε, μεγαλύτερο κίνδυνο. Οπωσδήποτε μια κατηγορία η οποία είναι πιο εκτεθειμένη είναι αυτή η ενδιάμεση οι οποίοι υπόσχονται εγγυημένες αποδόσεις. Αυτό ισχύει για κάποιες εταιρείε ε, ε, ασφαλιστικές ε, και για κάποια ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιδοτικά ταμεία. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι οπωσδήποτε η άνοδος των τιμών των ακινήτων που παρακολουθούμε σε κάποια μέρη της Ευρωζώνης, παρά το ότι δεν απέχουμε πολύ ακόμα από το να μιλήσουμε για κάποια φούσκα. Δηλαδή ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά δεν βλέπουμε κάποια έκρηξη της πίστης ε, και της μόχλευσης. Αλλά οπωσδήποτε τα χαμηλά επιτόκια είναι και πάλι γόνιμο έδαφος για μια συμπεριφορά η οποία επιβραβεύει την αναζήτηση αποδόσεων. Οπότε πρέπει να την παρακολουθούμε. Και τέλος θα πρέπει να σκεφτούμε την γενικότερη κερδοφορία του τομέα των τραπεζών και των ασφαλιών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε άλλα στοιχεία που αντισταθμίζουν. Την κατάσταση αυτή. Οπωσδήποτε υπάρχει ο αντίκτυπο στα κέρδη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά. Σα ευχαριστώ, κύριο Παπαδημούλη. Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη, επιτρέψαμε να σα ρωτήσω κάτι που φορά ιδιαίτερα στη χώρα μου την Ελλάδα σημείωσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, τη δήλωσή σας πριν από λίγο για τη σημαντική πρόδρο που έχει ε, σημειωθεί στην ελληνική οικονομία. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω και τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε από την πλευρά σας ε, για να ενισχυθεί αυτή η τάση και να σταθεροποιηθεί. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος που την είχατε θέσει ως προϋπόθεση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM αποδέσμευσε την περίφημη δόση. Η ερώτησή μου είναι πότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα αποφασίσει την άρση του waiver έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος του τραπεζικού δανεισμού και να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγματική ελληνική οικονομία. Να περιμένουμε μια τέτοια απόφαση αύριο. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά στη συμμετοχή και της Ελλάδας επιτέλους στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που όλοι θεωρούν ότι θα βοηθήσει την ταχύτερη επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη. Πότε εκτιμάτε ότι αυτό θα το αποφασίσετε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπό ποιε προϋποθέσεις και σε ποια έκταση. Και τέλος, το ενδεχόμενο μιας αναβολής ή μιας μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του τρίτου πυλώνα της τραπεζικής ενοποίησης που αφορά την πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων που σωστά το απέφιαστε και δεν το επιθυμείτε συνιστά ή όχι ένα συστημικό κίνδυνο για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Thank you. I mean, a bureaucratic answer to your question. Ευχαριστώ. Μια γραφειοκρατική απάντηση στην ερώτησή σας θα ήταν ότι μιλάμε τώρα για το Συμβουλίο Ιστημικής Σταθερότητας και όχι για την Κεντρική Τράπεζα, οπότε δεν συζητάμε την Ελλάδα στο Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας. Αλλά θα απαντήσω και πιο ουσιαστικά. Κοιτάξτε, τώρα που το ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας έχει λάβει την απόφαση του για τα προαπαιτούμενα και την ε, εκταμίευση, θα εξετάσουμε οπωσδήποτε ε, το θέμα του waiver και μπορεί να υπάρξει μια απόφαση η οποία θα οδηγήσει σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε επιλεξιμότητα για το πρόγραμμα ε, ποσοτικής ε, χαλάρωσης. Νομίζω έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχουν χρονικά όρια. Υπάρχουν όρια οπωσδήποτε στο ποιο ε, εκδίδει και βεβαίω υπάρχει και η αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα για την βιωσιμότητα του χρέους. Οπότε θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Φίλιπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για τον ε, κίνδυνο του να παραμείνουν πολύ χαμηλά τα επίπεδα του πληθωρισμού. Είδαμε τα επιτόκια, εδώ μιλάμε για χρηματοπιστωτική ε, σταθερότητα σε σχέση ε, με τον πληθωρισμό. Αυτό πώς θα επηρεάσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Χαμηλά επιτόκια τώρα. Αναφέρατε νωρίτερα πως ανεβαίνουν και οι επενδύσεις. Ανησυχώ όμως, διότι βλέπω πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες ε, χρησιμοποιούν πολύ χαμηλά επιτόκια ε, για να τροφοδοτηθούν ουσιαστικά. Και η εμπειρία δείχνει ότι δεν χρησιμοποιείται αξία ε, πολλές, από πολλές από αυτές τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που αντιθέτως ε, είναι αποτυχημένες ε, δραστηριότητες. Είναι χρήσιμο λοιπόν κάτι τέτοιο. Και τι σημαίνουν όλα αυτά από την πλευρά των συστημικών κινδύνων. Τέλος, θα ήθελα την άποψή σας για την ιδέα ότι ίσως ε, θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ζητώντας από τις ευρωπαϊκές τράπεζες να έχουν ένα χαρτοφυλάκιο δημόσιων χρεογράφων ε, τίτλων χρέων. Δηλαδή να μην συγκεντρώνεται ο κίνδυνο, παραδείγματο χάρη, από Ισπανικέ τράπεζε, στι Ισπανικέ τράπεζε, στο Ισπανικό χρέο. Αλλά κάθε τράπεζα να έχει ένα χαρτοφυλάκιο που ίσω να αντικατοπτρίζει και την κεφαλαϊκή δομή τη ΕΚΤΑ και αυτό νομίζω θα είχε μηδενικό, αξιολόγηση μηδενικού κινδύνου. Ποια είναι η άποψή σα, Απάντηση. πρώτη ερώτηση ήταν κατά πόσον ο χαμηλό πληθωρισμός επηρεάζει τον κίνδυνο. Ναι, φυσικά και τον επηρεάζει. Και ίσως τα νοικοκυριά εταιρείε, ίσως και ε, σε επίπεδο δημοσίου, οι αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από πάρα πολλά χρόνια, με βάση αυτό τώρα το ποσοστό του πληθωρισμού του 2%, τώρα έχουν, να αντιμετωπίσουν ένα χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού. Και αυτό σημαίνει υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για τα πραγματικά επιτόκια και μεγαλύτερο χρέος που επομίζονται. Εμείς περιμένουμε επιστροφή του πληθωρισμού στα επίπεδα του 2%. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τον πολύ χαμηλό πληθωρισμό για όλες ε, τις κατηγορίες ε, των ε, οφειλετών. Ιδίω όταν μιλάμε για κατηγορίε χρέου που ε, έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευση ε, πάρα πολύ παλιότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ε, κατά πόσον σχετίζεται αυτό ο πολύ χαμηλό πληθωρισμός και με τις κακέ κακές γενικώ μακροοικονομικέ μακροοικονομικές συνθήκες, αυτό είναι ένα άλλο παράγοντα κινδύνου που πραγματικά είναι διάχυτος και σημαντικός. Σε ό,τι αφορά τώρα εξαγορές και ε, συγχωνεύσεις αν πάμε πίσω στο 2006-2007 και στο 2005, οι όγκοι εξαγωγών και συγχωνεύσεων τότε ήταν πολύ μεγαλύτεροι από τη σήμερα. Και τα επιτόκια ήταν και ψηλότερα. Επομένως είναι σαφές ότι τα χαμηλά επιτόκια ενθαρρύνουν ε, τη χρηματοδότηση, το χρέος, ίσως λοιπόν ενθαρρύνουν και μοχλευμένες ε, συναλλαγές ε, M&A, συγχωνεύσεις, εξαγορές. Αλλά δεν νομίζω ότι περιμένουμε και καμιά τρομερή εξέλιξη σε σχέση με τα πρώτης κρίσης ε, επίπεδα. Δηλαδή δεν περιμένουμε, δεν παρατηρούμε συστημική αύξηση μόχλευσης τουλάχιστον στους, στον τομέα που μπορούμε να παρατηρήσουμε, δηλαδή τον τραπεζικό τομέα. Τρίτο ερώτημα. ένα νέο είδος περιουσιακού στοιχείου, ακίνδυνου εντελώς, χωρίς ρίσκο. Θα το συζητήσουμε αυτή τη βδομάδα στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Έχουμε ένα έγγραφο από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε. Δεν μιλάμε ακριβώς για το ίδιο κόνσεπτ με αυτό που είπατε εσείς, όμως ο στόχος, ο σκοπός μοιάζει. Μοιάζει κατά πολύ με αυτό που εσείς αναφέρατε. Έχει δημοσιευτεί αυτό το έγγραφο, λέει ο κ. Λάμπερτς. Θα δημοσιευτεί. Περιμένετε να δούμε πρώτα τι θα αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο για τη δημοσίευσή του. Πάντως περιμένουμε να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από αυτό το εγγράφο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σύντομες ερωτήσεις έχω. Πρώτα απ' όλα για τον κίνδυνο για τα ασφαλιστικά προϊόντα λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Γνωρίζουμε πως τα επιτόκια πρώτα απ' όλα τα χαμηλά βλάπτουν τους αποταμιευτές αλλά πλήττονται και άλλα προϊόντα, οι ασφάλειες ζωής και βεβαίως υποφέρουν και τα εταιρικά συνταξιοδοτικά ταμεία και τέλος οπωσδήποτε και οι ιδιωτικές ασφάλειες υγείας που έχουν και αυτές ένα κομμάτι αποταμίευσης το οποίο μειώνεται. Οπότε θα αυξηθούν οι εισφορές ε, είτε θα μειωθούν οι παροχές υγείας. Μήπως λοιπόν με την πολιτική σας μεταφέρετε τους κινδύνους από τον χρηματοπιστωτικό τομέα στον ιδιωτικό τομέα στην ασφάλεια υγείας και ζωής ε, από, τις, ε, από τους ιδιοκτήτες των τραπεζών, δηλαδή στους ηλικιωμένους και τους ασθενείς. Και δεύτερη μου ερώτηση αφορά τα πρακτικά. 10 Μαΐου 2016 τουλάχιστον αναφέρεται στο, έτσι, στο site της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας μιλεί, απαντήσατε στο θέμα ε, της μετάβασης από τα επιτόκια σε μη συμβατικά μέσα και ερωτηθήκατε εάν θεωρητικά θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται το λεγόμενο χρήμα με το ελικόπτερο όπως λέγεται. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Το είπατε όντως αυτό ή γράφει λάθος πράγματα η σελίδα της ε, τράπεζας. Και τέλος για τον κίνδυνο λόγω του χαμηλού πληθωρισμού ο πρόεδρος διακόπτη. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, αλλά έχουμε και ψηφοφορία μετά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πρώτη ερώτηση αφορά τον κίνδυνο για τον κλάδο των ασφαλιών. Οπωσδήποτε παρακολουθούμε τον κίνδυνο αυτόν πάρα πολύ προσεκτικά και ειδικά τον κίνδυνο που πηγάζει από τα χαμηλά επιτόκια. Και αυτός ο κίνδυνος βεβαίως αφορά κάποια συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα, ειδικά της ασφαλής ζωής που προσφέρουν ε, κάποιες υψηλές εγγυημένες αποδόσεις. Να σας πω το εξή όμως, το είπα και πριν. Οι είχαν 8-9 ε, χρόνια μηδενικά επιτόκια και δεν άκουγε κανείς τέτοια παράπονα, αυτά τα οποία ακούμε από την Ευρωζώνη ή τμήματα της Ευρωζώνης. Δεν ακούγαμε πως θα επηρεαστεί η υγεία από τα μηδενικά επιτόκια. Και η υγεία εκεί είναι ε, και ήταν ε, κατά κανόνα ε, ιδιωτική. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να επηρεαστεί η υγεία από τα χαμηλά επιτόκια στην Ευρωζώνη, αλλά να επανέλθω στις ασφαλιστικές εταιρείες. Λοιπόν, η οδηγία για τη φερικαιότητα 2, η οποία φέρνει τον υπολογισμό της φερικαιότητας πιο κοντά σε αυτά τα οποία έχει η αγορά, θα αυξήσει και την διαφάνεια. Οπότε, στη μετάβαση προς αυτό το καθεστώς, οι εταιρείε μπορούν να έρθουν να χρησιμοποιήσουν μεταβατικά μέτρα τα επόμενα 16 χρόνια και έτσι θα αποφευχθούν η δραματικές αλλαγές στη μετάβαση στο νέο καθεστώς. Επίσης, αναλύσαμε τον δυνητικό κίνδυνο που προκύπτει από αυτές τις δραστηριότητες και αυτά δημοσιεύτηκαν το τέλος του 2015, τέλος για τα λεφτά τα οποία θα ρίχναμε το ελικόπτερο. Δεν συζητήθηκε αυτό ποτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπερναρ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρος επικεφαλής λοιπόν του Συμβουλίου Συντημικού Κινδύνου για πέντε χρόνια διερωτώνται πολύ πόσο αποτελεσματικός είναι αυτός ο θεσμός και ποιος είναι ο ρόλος. Δημιουργήθηκε το 2004 ο μηχανισμός Ενίας εποπτεία, το SSM, και απέσυρε τα ουσιαστικά τη χρησιμότητα του Συμβουλίου ε, Κινδύνου, αυτού του Συντημικού κινδύνου. Δεν ακούσαμε στην αρχή του έτους να μας αναφέρεστε όσον αφορά τα, τα κοκό της Deutsche Bank και τα διάφορα χρεόγραφα. Ούτε προβλέψατε, ούτε αναλύσατε των προτέρων της ε, βεβαιότητας όσον αφορά την Deutsche Bank. Οι περισσότερε χρηματοπιστωτικέ κρίσει ξεκίνησαν από ανισορροπίε στη χρηματοπιστωτική αγορά, αλλά εξακολουθεί το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου να αγνοεί τι συστημικού κινδύνου τη αγορά. Παραδείγματο χάρη, η δημιουργία μια αποζημίωση των συναλλαγών των παραγωγών χάρη ε, στον έλεγχο τη αγορά Εκεί συγκεντρώνεται ο συστημικός κίνδυνος των υποδομών. Αυτό μπορούσε να γίνει μια ορολογική βόμβα. Το επεξεργάζεται το θέμα αυτό. Ποιον άξονα ακολουθείτε στον προβληματισμό. Επιβεβαιώνεται μετά τις πληροφορίες η μεταφορά αρμοδιοτήτων από των κοκκίνων των δανείων από τι εθνικέ Τράπεζες προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ για την απάντησή σα εκ των προτέρων. Thank you. Απάντηση, ευχαριστώ. Να πω μερικά λόγια για το ρόλο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου εξετώντας το όλο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να θυγραμμίσουμε διαδικασίες και τη χρήση διαφόρων εργαλείων, ούτως ώστε να περιορίσουμε ενδεχομένως ε, προβλήματα και να αυξήσουμε την αντοχή ε, του χρηματοστικού συστήματος και την ισορροπία αυτού. Το περιεχόμενο των νομοδοτήσεων ε, του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, διότι δεν λαμβάνουμε αποφάσεις ως φορέας, αλλά είμαστε φορέας που γνωμοδοτεί και εκδίδει συστάσεις και προειδοποίησεις. Αυτή η γνωμοδότηση παρόλα αυτά αντικατοπτρίζει τη μεταμόρφωση του οικονομικού τοπίου, του οποίου υπήρξαμε μάρτυρες τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή της κεφαλογικής ενιαίας αγοράς για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η επέκταση του μετραπεζικού τμήματος του τομέα ή τα προβλήματα δημιουργούνται από τα χαμηλά επιτόκια ζητούν προοπτική που δημιουργείται και δεν περιορίζεται όμως αποκλειστικά στο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, ενώ το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ήδη έχει δώσει στον Ευρωπαίο Νομοθέτη απόψεις σχετικά με δεχόμενες επιλογές και αναθεωρήσεις που θα χρειαζόταν στα πλαίσια ε, των αυματικών αναθεωρήσεων που έγινε το 2014, επίσης προβληματιζόμεθα επί πολιτικών που ήδη έχουν γίνει στον τομέα εκτός ε, τραπεζικού. Πρέπει να περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το, για το πεδίο εφαρμογή της ε, αναθεωρήσεως, το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων και το τελικό αποτέλεσμα της νομοθετικής προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα. Σας ευχαριστώ. Του ELA, για το θέμα του ELA, μπορείτε να απαντήσετε, τις αρμοδιότητες του ELA. Ε, δεν θα απαντήσει το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου επ' αυτού, δεν αρμοδιότητά μας. Θα πρέπει να ομοδοποιήσουμε τις τελευταίες ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη λόγω χρονικών περιορισμών. Καταρχάς ο κύριος Ζάλμπα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ντράγκη, Ομιλώ εκ μέρους της Εύα Παούλοβα, της αγαπητής συναδέλφου. Θα διαβάσω την ερώτηση, μάλλον του κυρίου Παλόβα. Συγχαρητήρια για τα πρώτα έτη των εργασιών του Συμβουλίου σας που λειτουργήσε με συνέπεια, αλλάζοντας το, το ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο. Αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα και προκλήσεις στα πλαίσια της ολοκληρώσης τραπεζικής ενώσεως. Η μείωση του κινδύνου, του συστημικού, είναι ένας από τους στόχους και τα προβλήματα. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων κρούσεων. δεν υπάρχουν σαφείς συστάσεις πολιτικής όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου. Εν τη απουσία του ενδεδειγμένου μηχανισμού, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προχωρήσει όσον αφορά το σχέδιο ασφαλίσεως των καταθέσεων. Ποιο θα είναι τα βασικά στοιχεία νέου κανονισμού για τις εκθέσεις των κρατικών ομολόγων και πώς μπορούμε να αποφύγουμε ασύμετρη κατανομή των δαπανών στις τράπεζες ή στους εκδότες ε, τίτλων στις διάφορες χώρες. Άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μακροοικονομικό που ενθαρρύνει το μη τραπεζικό τομέα Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι έχει δρομολογική ήδη ε, η προσπάθεια όσον αφορά αυτά τα εργαλεία στο Συμβούλιο σας, στο μη τραπεζικό τομέα. Ποιο θα είναι το σημαντικότερο στοιχείο ενός νέου μακροοικονομικού πλαισίου που θα αποφεύγει τον κίνδυνο στο μη τραπεζικό τομέα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, συζητήθηκε και στο Συμβούλιο. Εδώ συζητούμε τη ρύθμιση για τη δημιουργία τετλοποιήσεων STS, ε, απλίες, ε, διαφανείς, ε, τυποποιημένες. Η ρύθμιση ως ισχύει αυτή τη στιγμή ε, περιλαμβάνει ένα ποσοστό διακράτησης αυτών των τιτλοποίησεων τάξης του 5% ε, στους τραπεζικούς ισολογισμούς και η πρόταση του εισηγητή της Επιτροπής μας ενός ε, συντρόφου από τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Πολ Τάγκ είναι να ανέβει στο 20% αυτό το ποσοστό. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι τα μέτρα κεφαλαικών απαιτήσεων είναι μέτρα μικροπροληπτικού χαρακτήρα. Και επομένω ρωτώ, με δεδομένο ότι αυτές οι τιτλοποιήσεις ε, αγοράζονται από μη τραπεζικούς φορείς. Και επειδή ένας από τους στόχους είναι η σταθεροποίηση και η ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα, του shadow banking, δεν θα ήταν σκόπιμο τελικά αυτές, αυτή η διακράτηση της πίστης να εξαρτηθεί και από τη θέση στον κύκλο. Δηλαδή αν έχουμε ένα boom στο shadow banking και θέλουμε να το ελέγξουμε αυτό το shadow banking, να μπορούμε να αυξάνουμε αυτό το ποσοστό διακράτηση και να μειώνουμε αντίστοιχα. Δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τελικά αυτό ως στοιχείο μακροπροληπτικού χαρακτήρα για να παρακολουθούμε, να επιτηρούμε και να ελέγχουμε, το, να συγκρατούμε μάλλον το σκιό τραπεζικό τομέα. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτός ένας ε, δρόμος για να βελτιώσουμε το συστημικό κίνδυνο του shadow banking. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Το πρώτο σας ερώτημα αφορούσε το έντις. Δεν μπορούμε όμως ε, να το, πούμε, να το συζητήσουμε. Το ξανάπαμε. Το, η ΕΚΤΑ θεωρεί ότι είναι ο τρίτος πυλώνας για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, το ΕΝΤΙΣ. Ε, πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση σίγουρα για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι έχουν τώρα ανασταλεί διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να βρεθεί ένα συμβιβασμός μεταξύ του επιμερισμού κινδύνων ε, και της εξάλληψης κινδύνων, de-risking, και θα πρέπει να δούμε και το χρονοδιάγραμμα όλων των δράσεων. Ουσιαστικά ε, είναι οι διόψεις ε, του νομίσματος αυτά, το de-risking και το risk sharing. Θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, την έκθεση ε, στο δημοσιογράφο αυτό που είπατε. Δημοσιεύθηκε για τα sovereign exposures τον προηγούμενο Μάρτιο ε, μία έκθεση για τα κρατικά αυτά ομόλογα και είπαμε ότι χρήζουν προτιμησιακής μεταχείρισης σε σχέση με τερικά ομόλογα ή άλλα και είδαμε δεν είναι το, τα κρατικά ομόλογα ε, απαλλαγμένα από κινδύνους. Το είδαμε και με, το δημόσιο χρέος και τη σχετική κρίση. Επομένως υπάρχει σύνδεσμος, το ξέρουμε. Μεταξύ κρατικού χρέους και τραπεζών και αυτό στο σύνδεσμος ήταν και ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο τραπεζικός τομέας. Και επηρέασε αρνητικά μεταξύ άλλων και τους διάβλους μεταδόσεις νομισματικής πολιτικής. Το Συμβούλιο Συντημικού Κινδύνου υποστηρίζει τα μέτρα για τη μετρίαση αυτών των κινδύνων, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια μεταβατική φάση, phasing in, και πρέπει να υπάρχει και συμμόρφωση με τη Βασιλεία Δηλαδή οποιαδήποτε αξιολόγηση και οποιαδήποτε αλλαγή στη μεταχείριση αυτών των κρατικών ομολόγων που τα έχουν στη κρατοχή τους οι τράπεζες θα πρέπει να ενταχθεί σε μια γενικότερη διαπραγμάτευση και δεν θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφασιστεί μόνο σε επίπεδο ένωσης ή ευρωζώνης που είναι ακόμα και πιο δύσκολο να το καταλάβει κανείς στην έκθεση. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το Συμβούλιο Συντημικού Κινδύνου έχει μια ανάλυση 70 σελίδων για μια σειρά από επιλογές πολιτικής και στην έκθεση καταγράφονται αυτές οι επιλογές μεταρρύθμιση κεφαλικών απαιτήσεων για τις τράπεζες σε 1, κίνητρα πολιτικής για μεγαλύτερη διαφοροποίηση, μεγαλύτερη ε, αποκάλυψη, σχετικοί κανόνες κτλ. Άρα είναι εκτεταμένη έκθεση διεξοδική, βλέπετε υπέρ και τα κατά των διαφόρων ε, επιλογών δεν τοποθετείται όμως για τη σχετική τα υπέρ και τα κατά αυτών των επιλογών. Απλά τα αναφέρει. Και όλα αυτά ε, συζητούνται και σε επίπεδο EFC, ε, σε επίπεδο της Επιτροπής της Βασιλείας, της ΕΚΤΑ και από το Συμβούλιο στην Κινδυνού συζητούνται όλα αυτά. Κάποια στιγμή τέλος πάντων όλος αυτός ο συλλογικός προβληματισμός ε, θα καταλήξει σε μια άποψη που πιστεύουμε ότι θα βρίσκει σύμφωνο σε όλους τους συμμετέχοντες. Το άλλο σας ερώτημα αφορούσε τον μη τραπεζικό τομέα και τα εργαλεία μακροπροληπτικού χαρακτήρα για τον μη τραπεζικό τομέα. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε κάποια από αυτά τα εργαλεία. Δεν θα είναι σίγουρα πλήρης αυτός ο κατάλογος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι εργαλεία τα οποία θα αντιμετωπίζουν αντιστοιχίες ρευστότητα, επενδυτικά ταμεία κτλ. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μέσα εργαλεία τα οποία θα αντιμετωπίζουν την προκυκλικότητα, αρχικά περιθώρια ή κούρεμα ε, στις διάφορες συναλλαγές, ε, σε χρεόγραφα και σε παράγωγα. Όπως γνωρίζετε, το έχει αναλάβει τη μακροπροληπτική εποπτεία συνολικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα έχει ηγετικό ρόλο για την ανάπτυξη της στρατηγικής μιας πολιτικής μακροπροληπτικού χαρακτήρα και θα αντιμετωπίζουμε κινδύνους πέραν και του τραπεζικού τομέα. Σίγουρα θα συνεργαστούμε με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα ή FSB που έχει ξεκινήσει τις εργασίες του ήδη εδώ και κάποιο καιρό. Σε ό,τι αφορά τις τυπλοποιήσεις TST, απλές διαφανείς τυποποιημένες, είμαστε υπέρ της πρότασης Κομισιόν. Στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση στην αγορά πίσω, που μέχρι στιγμής είναι περιορισμένη. Λόγω και των πολύ απλών, χαλαρών, επεκτατικών όρων χρηματοδότησης και το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να πω ότι δεν οδηγεί σε μια τέτοια θετική εξέλιξη. Γι' αυτό και η πρόταση Κομισιόν μας βρίσκει σύμφωνους. Συμφωνούμε, παραλαμβάνω, με την πρόταση Κομισιόν και για τα τέλεια κράτησης κεφαλαιακά κτλ. Ο βασικός στόχος για να έχουμε αυτή την απλή διαφανή τυποποιημένη τιτλοποίηση είναι να έχουμε κεφαλαιακές χρεώσεις που δεν θα είναι ίδιες με τις μη απλές ε, διαφανείς και τυποποιημένες ε, τιτλοποίησεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κατάσταση είναι απότοκο της κατάστασης που προέκυψε μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, όπου όλες τις τετλοποιήσεις ε, που αγοράζονταν σας ΣΥΠΑ και, στις, ε, και στην Ένωση αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Αλλά είχαμε ένα default rate που ήταν το 1 δέκατο στην Ένωση σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και τα, οι τίτλοποιήσεις μας τιμολογούνταν ε, εύκολα, ήταν ευανάγνωστες, ήταν διαφανείς, εγκρίναμε τον ίδιο κανονισμό. Η Κομισιόν λοιπόν προτείνει ε, κάτι που θα διορθώσει αυτές τις διαφορές. Τώρα αυτή η διακράτηση, αυτή, αυτό το ποσοστό λέτε εσείς θα πρέπει να αλλάζει με, ανάλογα με τον αγοραστή. Θα το σκεφτούμε. Νομίζω ότι είναι ζήτημα που αφορά πιο πολύ την προστασία των καταναλωτών και όχι τόσο το βέλτιστο σχεδιασμό ενό ε, χρηματοπιστωτικού πρότυπου, αλλά το σκεφτούμε. Thank you very much uh, to President Draghi. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Ντράγκη. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σημαντικότητα τη συζήτηση στο δεύτερο τμήμα του νομισματικού αυτού διαλόγου. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να υπενθυμίσουμε ότι η είναι αποφάσισε όσον αφορά το κρατικό χρέος, να μην υπάρχει εμπροστοβαρής αντιμετώπιση και να αναμένουμε τη Βασιλεία. Συνετή απόφαση που ταιριάζει με αυτά που ψηφίσαμε, θα επανέλθουμε από αυτόν, αφού διαβάσουμε τις νέες μελέτες και τις ε, διάφορες επιλογές που μελετά το Συμβούλιο ε, του Συστημικού Κινδύνου, διακοπή δύο λεπτών και μετά θα ψηφίσουμε. We have to start voting, dear colleagues. Ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, συναδελφοί. Ήδη έχει ανακοινωθεί πως θα υπάρξει μια ονομοδότηση τη μειοψηφία. Έχει αποσταλεί στην γραμματεία. Λοιπόν, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Λοιπόν, ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Συμβαστική α υπέρ. Κατά εποχές δεκτή. Συμβαστική β υπέρ κατά εποχές δεκτή συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχες δεκτή τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή ε υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική G υπέρ σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.49 υπέρ κατά αποχές δεκτή Άι, μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 116 υπέρ κατά αποχές δεκτή 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική αι α με προφορική τοπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική J υπέρ κατά αποχές δεκτή 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική K υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική μη υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική νη υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 133 υπέρ. Κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε την 133. Άρχεται η 133. Πέρας απορρίπτεται ο μικρόν υπέρ κατά αποχές δεκτή π υπέρ κατά αποχές δεκτή Q υπέρ κατά αποχές δεκτή Q α υπέρ κατά αποχές δεκτή R υπέρ κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή S υπέρ κατά αποχές δεκτή 153 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 158 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές κατά αποχές να την απαλληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 158. Προφορική τροπολογία, ναι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν πενήντα Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συναστική τάφ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 168 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική U υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική V υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται W υπέρ κατά αποχές δεκτή 198 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική X υπέρ σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές δεκτή Z υπέρ κατά αποχές δεκτή αλφα αλφα υπέρ κατά αποχές δεκτή 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 226 υπέρ κατά αποχές δεκτή 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ΕΑΒ υπέρ κατά αποχές δεκτή AC ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.43 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή προτείνω να ψηφίσουμε όλες μαζί την 1 έως 10 της Επιτροπής Πολιτισμού συμφωνείτε όχι όχι κουλτ 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, τη λογική σκέψη 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή 3α με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 έως 7 μαζί τη λογική σκέψη κατά αποχές δεκτές 7α προφορική τροπολογία υπέρ κατά ε, δεκτή από το 8 μέχρι και την 15 όλες μαζί συμφωνείτε υπέρ κατά αποχές δεκτές 15α με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 15β με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο 17 και 18 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική αε υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική AF υπέρ κατά αποχές δεκτή AG υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά ΕΛΚ υπέρ δεκτή συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές δεκτή ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας 46 υπέρ 8 κατά Δύο αποχές συγχαρητήρια Συγχαρητήρια κύριε Κάρας. Ναι, είπαμε ότι έχουμε λάβει την έκθεση της μειοψίας που είπε Βαλεϊγκούε, το είπα στην αρχή. Επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 27 Ιουνίου από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεδρίαση.